θεωρούσαμε ότι θα τηρούν τα, ε, το δίκαιο που έχουν ψηφίσει οι ίδιοι. Και όταν ένας οργανισμός που είναι η Ευρωπόλ που υπόκειται στο κοινοτικό δίκαιο θεωρεί ότι δεν τη δεσμεύει και συγκεκριμένα εννοώ το άρθρο 4 της συμφωνίας, ε, τότε ορισμένα πράγματα πάνε στραβά. Δηλαδή, τίθεται το ερώτημα και όχι μόνο σε ποιο βαθμό τέτοιου είδους συμφωνίες στο μέλλον μπορούν να ευσταθούν και να έχουν νόημα, αλλά και πού είναι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου και κυρίως της Επιτροπής μας εδώ, ότι ε, ε, θα τηρείται αυτή η συμφωνία, την οποία εμείς εγκρίναμε. Τι θα πούμε στους πολίτες μας. Όταν ψηφίζουμε κάτι, όταν ε, αποφασίζουμε κάτι, θα πρέπει να εφαρμόζεται με τον τρόπο που ψηφίστηκε. Και ακριβώς αυτό δεν συνέβη με το θέμα του SWIFT. Το άρθρο 4 λέει ότι οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο στενές. Η δική σας έκθεση λέει το αντίθετο, ότι δεν μπορέσατε να τα ελέγξετε αυτά γιατί δεν είχατε πρόσβαση στα έγγραφα. Επίσης, λέει η συμφωνία ότι θα πρέπει αυτά να είναι γραπτά. Άρα πρέπει να έχουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Και τώρα ερχόμαστε και διαβάζουμε ότι γίνονται όλα προφορικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τίποτα δεν κατοχυρώνεται στο χαρτί. Μα δεν κάναμε μια συμφωνία για να παίξουμε πόκα είναι ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα των πολιτών μας. Δεν λέω, είναι θεμητός και αξιόλογος ο στόχος και ο σκοπός, αλλά δεν μπορούμε να αποφασίζουμε τέτοια πράγματα, να δίνουμε το ok, τις ευλογίες μας, να μας δίνουν διαβεβαιώσεις ότι όλα θα είναι ε, κανονικά και στο τέλος να μην τηρούνται. Αυτό δεν είναι υπεύθυνη νομοθεσία και επίσης δεν είναι νομοθεσία που να αποκαθιστά την αξιοπιστία των πολιτών ε, και της πολιτικής στα μάτια των πολιτών μάλλον και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ε, λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Η έκθεση σας είναι 5-6 σελίδες και τα πιο συχνά που διάβασα εκεί, οι πιο συχνές λέξεις ήταν impossible ή ότι ε, κατέστη αδύνατο κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται αυτό, δεν θέλει αυτό ο νομοθέτης και αυτός που κάνει τις συμφωνίες. Τώρα δεν ξέρω τι να προτείνω. Ο κύριος ε, Wainwright πώς ε, δικαιολογείται, πώς απολογείται ως Διευθυντής Ευρωπόλ, γιατί δεν μπορεί να μας λένε ότι είναι απόρριτα, εμπιστευτικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και δεν τηρείται η συμφωνία, αλλά... Ε, ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη, και εδώ δεν αφορά την Ευρωπόλ, δεν ανταποκρίνονται ε, στην υποχρέωση που έχουν να ε, απαντούν οι επόπτες προσωπικών δεδομένων σε ερωτήσεις των πολιτών. Εγώ ρώτησα ιδία πρωτοβουλία το γερμανό επόπτη προσωπικών δεδομένων, αν μπορούν να μου δώσουν πληροφορίε ποια στοιχεία έχουν διαβεβάσει για μένα, για τι δικέ μα συναλλαγέ στι ΗΠΑ. Μετά από έξι μήνε, η απάντηση που ήρθε ήταν αδύνατο. Δεν μπορούμε να σα πούμε ποιε συναλλαγέ σα. Και μάλιστα με αποθαρρύνουν να ρωτήσω γιατί οι ΗΠΑ δεν θέλανε μόνο τα στοιχεία τη ταυτότητά μου, αλλά και τον αριθμό λογαριασμού μου. Ε, τι να το κάνουμε όλο αυτό, πού είναι η προστασία των δεδομένων. Πρώτα με απογυμνώνουν και μετά δεν μου λένε και τι ξέρουν για μένα. Και χρειάστηκαν μισό χρόνο για να μου πούνε όχι και να μου πούνε ότι είναι αδύνατο. Δεν ήταν σε θέση να μου πούνε εάν ε, έδωσαν στοιχεία, ποια στοιχεία έδωσαν για μένα και ποιος τα έχει στα χέρια του. Μετά από έξι μήνες SWIFT. Συμπέρασμα. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Θα συνεχιστεί η διακατάσταση χωρίς να έχουμε ούτε ίχνος προστασία των πολιτών, προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, με εφαρμογή όλων αυτών. Τότε τι θέλαμε όλη αυτή τη συμφωνία. Α το κανονίζαμε μεταξύ του τα κράτη, αφού έτσι κι αλλιώ δεν παίρνουμε σοβαρά υπόψη αυτά που αποφασίζει το Κοινοβούλιο. Και παρακαλώ να αναρωτηθεί κάθε πολιτική ομάδα πόσο σοβαρά μα παίρνουν υπόψη όταν πρόκειται για την επιβολή και την εφαρμογή του νόμου. Προσωπικά περιμένω να έρθει ο κύριος Γουένραϊτ να απολογηθεί γιατί δεν τηρήθηκε το άρθρο 4 της συμφωνίας και ελπίζω να έχω απαντήσεις στην έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε συστάσεις στη σελίδα 6 της έκθεσής σας πάρα πολύ χρήσιμες και ωφέλιμες και θεωρώ σκόπιμο να σκεφτούμε μέχρι και αναστολή της συμφωνίας. Αν δούμε ότι από ό,τι φαίνεται δεν τηρούνται, αγνοούνται αυτές οι ρυθμίσεις ασφαλείας. Όταν είπαμε εμεί το OK για αυτή τη συμφωνία, δεν είχαμε υπόψη μα ότι θα συμβούν τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αλβάρο. Ο κύριος Μπουσουτήλ από τους ε, συντονιστές μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Μία για τη διαδικασία, η δεύτερη επί της ουσίας. Ας με την διαδικασία. Νομίζω είναι λίγο παράξενο ότι εδώ μιλάμε για μια έρευνα η οποία έγινε ε, το Νοέμβριο, μια έκθεση που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο και ε, μια έκθεση τουλάχιστον ε, ένα ανακοινωθέν τύπου που φτάνει σε εμά το Μάρτιο. Γιατί μπορείτε να μου εξηγήσετε, έπρεπε να περιμένουμε τόσο πολύ να λάβουμε να, να μας δοθεί αυτή η ενημέρωση. Δεύτερον, επί της ουσίας. Καταλαβαίνω ότι τα συμπεράσματα της ΚΕΑ είναι ότι είναι αζύνατο να αξιολογήσετε εάν τα δεδομένα τα οποία μεταφέρθηκαν, τα οποία διαβιβάστηκαν, ήταν αναγκαία να διαβιβαστούν και ήταν και ε, τα σωστά. Αυτό δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι γίνεται, διότι από πέρσι ε, και εγώ και οι συνάδελφοι είχαμε πει ότι δεν είμαστε διόλου ευχαριστημένοι με αυτή τη μοναδική ε, ρήτρα ασφαλείας που λέει ότι η Europol είναι ο μόνος ελεγκτικός φορέας που θα ελέγχει αυτές τις διαβιβάσεις δεδομένων. Εμείς ζητήσαμε μια συμπληρωματική ρήτρα ασφάλειας, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα, θα είναι στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ως μόνη αρμοδιότητα θα έχει την παρακολούθηση της διαβίβασης αυτών των ας πούμε στοιχείων των δεδομένων στο μαύρο κουτί. Η Europol δεν μπορούσε ποτέ να έχει τον έλεγχο κάθε μεμονωμένου στοιχείου, δεδομένου. Έστελνε δεδομένα χίδιν, ας πούμε, μέσα στο μαύρο κουτί και έτσι χανόταν. Ε, τα, τα, οι λεπτο, χανόντουσαν οι λεπτομέρειες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι υπεύθυνο να εξετάζει αιτήματα για, την, για λεπτομερείς ε, ε, όταν ε, προκύπτει με τέτοια περίπτωση από πλευράς Europol προς τις Αμερικανικές Αρχές. Εγώ πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι ικανοποιητική από πλευράς Europol. Πιστεύω όμως ότι η κοινή εποπτική αρχή λειτουργεί σωστά, κάνει σωστά την εργασία της και τέλος Κατά λίγο είχαμε υιοθετήσει δύο άλλες ρήτρε ασφαλείας. Η πρώτη, επειδή ακριβώς δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με αυτήν την μετα... Ε, διαβίβαση στοιχείων χίδιν, είχαμε πει εδώ στο Κοινοβούλιο και χάρη αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαμε πιέσει να γίνει ένα ευρωπαϊκό κοινοτικό TFTP για να σταματήσουμε αυτήν την ανεξέλεγκτη διαβίβαση στοιχείων. Σας θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε πού βρισκόμαστε σε αυτήν την προ... για την πρόσφαση ενό κοινοτικού TFTP. Και δεύτερη ρήτρα ασφαλείας είχαμε ζητήσει μια γενική, γενική ε, έκθεση η οποία θα αξιολογεί όχι μόνο το ρόλο της Ευρωπόλ μέσα στο TFTP, αλλά γενικά μέσα στην ευρύτερη συμφωνία. Ελπίζω αυτή η αναθεώρηση, η έκθεση αναθεώρησης να έρθει σε εμά ε, σύντομα και προσβλέπω στην ενημέρωση από πλευράς Επιτρόπου. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να τονίσω εκ μέρους της ομάδας μου ορισμένα σημεία που ελέξησαν στην αρχή-αρχή της συζήτησης θέλω να σας εκφράσω και εγώ τις επιφυλάξεις μας, ως ομάδα δηλαδή, όπως το είπε και ο κύριος Αλβάρο και άλλοι προλαλήσαντες, ότι η έξεση της ΚΕΑ αναπόφευκτα θα έλεγε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ευρωπόλ να συμμορφωθεί σε αυτές τις ε, ισχυρότατες απαιτήσει του, Υπουργείου, του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Ε, είναι πολύ γενικές και ασεφείς ε, η, μαζική διαβίβαση δεδομένων υπό τη συμφωνία SWIFT. δυστυχώς επαλυσσεύονται οι αρχικές επιφυλάξεις που είχαμε. Από πλευράς δικής μου ομάδας είχαμε ζητήσει, ε, μείναμε μία ε, επεξήγηση του άρθρου 4 ε, για να δούμε πώς θα γίνεται σωστά η επαλήθευση των δεδομένων. Είχαμε πει ότι τα υπάρχει ασφαλώς ε, ανάγκη στα δεδομένα αυτά, ιδίως για την τρομοκρατία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Europol, να οι απαιτήσει για διαβίβαση στοιχείων να είναι όσο το δυνατόν ε, πιο λίγες, ελάχιστες από την υπεραλληλαντική πλευρά. Τώρα προφορικές ενημερώσεις και προφορική συμφωνία κυριών δεν καταλαβαίνω τι σοϊ πράγματα είναι αυτά. Αυτή είναι μια πραγματικά πολύ παράξενη διαδικασία. Η προφορική παροχή δεδομένων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω ε, την ε, διαβίβαση συμπληρωματικών, ε, συμπληρωματικής τεκμηρίωσης προς την Europol και την εξέβρεση μιας ικανοποιητικής λύσης για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων της Europol. Η Επιτροπή οποία έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η επίλυση αυτού του προβλήματος αποτελεί μέρος των εργασιών της Επιτροπής και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα βασισμένο στην κοινοτική νομοθεσία, στην ε, νομοθεσία της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να μην λειτουργεί το πλαίσιο αυτό, όλη η διαδικασία διαβίβαση στοιχείων με ασαφή ε, ε, κριτήρια και διατάξεις, να είναι συγκεκριμένο και ασφαλές. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων, κυρία Α, λάθος, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος, δεν σας είχα στο, στη λίστα μου. Θα, θα είμαι πολύ σύντομη λέει η κυρία Βέμπερ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το πώς εγκρίθηκε αυτή η έκθεση. Εγώ έδωσα μάχη και ίσως έκανα λάθος, αλλά τέλος πάντων η ερώτησή μου τώρα αφορά την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στην Europol σαν ευρωπαϊκός οργανισμός, ευρωπαϊκή υπηρεσία, την οποία εγώ ήθελα να υποστηρίξω, να οφείλω να ομολογήσω ότι τώρα βρίσκομαι, είμαι κάπως μπερδεμένη, δεν ξέρω ποιο δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσω. Ποιο, ποιο είναι το συμβούλιο στο οποίο ο διευθυντής της Europol ε, είναι υπόλογος. Εγώ κατάλαβα ότι εσείς είσαστε υπεύθυνος ε, το γεγονός ότι θα αρνήθηκε η πρόσβαση. Εδώ ο Διευθυντής ήρθε πριν από μερικές εβδομάδες, ε, μας είπε για τους Αμερικανούς, ε, γιατί ότι είναι στο γραφείο, ε, ούτως ή άλλως τους Αμερικανούς βλέπουμε παντού. Όμως η Europol διαβιβάζει στοιχεία με βάση τις προφορικές συζητήσεις, να κρύψει ε, να κρύψει ένα τέτοιο στοιχείο από τους βουλευτές, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι τεράστιο λάθος. Θα τον καλέσουμε ξανά και θα ήθελα να έχουμε και την έκθεση, ήθελα τότε να, ε, να είχα την έκθεσή σας, ε, αλλά δεν την είχαμε, αλλά τέλος πάντων θα τον καλέσουμε. Θεσμικά όμως, πώς θέλετε εσείς να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος ο κύριος Άλμπραχτα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς σας συμφωνώ ότι προφανώς είναι καλύτερα ο κύριος Μπρέινράιτ να απαντήσει άμεσα σε αυτές τις ερωτήσεις, γιατί εμείς σαν κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγχουμε την Europol και αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση και η προσωπική μου άποψη αλλά και η άποψη των πρασίνων ήταν σαφές από το καλοκαίρι ότι η στάση αυτή δεν ευθυγραμμίζεται δεν ευθυγραμμίζεται με τις βασικές μας αρχές. Προφανώς αυτές οι μεταβιβάσεις στοιχείων και δεδομένων είναι ακριβώς το αντικείμενο για το οποίο μας ασκείται κριτική. Δεν μπορεί να έχουμε ένα, ένα άτομο δεν μπορούμε μάλλον να κατηγορούμε ε, ένα άτομο και μόνο, αλλά θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένες πληροφορίες, ποια είναι τα στοιχεία, ποια είναι τα δεδομένα τα οποία επεξεργαστήκαμε κτλ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις ε, ε, αρχές μας, με τις συνταγματικές αρχές ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξάγει κάποια συμπεράσματα. Εδώ υπάρχουν όντως σαφέστατες παραβιάσεις και κανένα δικαστήριο δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε κανένα, ούτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ούτε κανένα άλλο, δεν θα ε, δώσει το πράσινο φως θα τονίσει το γεγονός ότι δεν ευθυγραμμίζεται η συμφωνία αυτή με, την, ε, ε, με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς δημιουργήσαμε μόνοι μας. Δεν, ευθύνεται η δεν ευθύνονται οι Ηνωμένε Πολιτείε. άρα θα πρέπει και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δούμε τι ακριβώς δεχόμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν συνάδει με την νομοθεσία μας και τις θεμελιώδεις αρχές. Ο κύριος Κίκο. Πρόεδρε, έχετε απόλυτο δίκαιο όταν αναφερθήκατε στην ε, συντομία κάποιων παρεμβάσεων. Ε, με εκπλήστο γεγονό ότι δεν υπήρχαν ε, πολλά πράγματα να πούμε. Τέλος πάντων, εγώ υποστήριζα πάντοτε αυτή τη συμφωνία και ξέρω ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν ασκήσει κριτική και έχουν επιτεθεί στις Ηνωμένες ε, για τους στόχους τους και τους σκοπούς τους. Αλλά ειλικρινά νομίζω ότι έχουμε κάνει λάθος στόχο εδώ. Όλη αυτή η κατάσταση προφανώς ε, είναι ε, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εγώ ενέκρινα, εγώ ξέρετε, το ξέρετε όλοι ότι ήμουνα υπέρ αυτής της συμφωνίας, γιατί ακριβώς θεωρούσα ότι είχαμε επαρκείς ρήτρε διασφάλισης ε, για τα δεδομένα που αφορούν τους πολίτες μας και αυτά τα οποία άκουσα τώρα ε, με απογοητεύουν, διότι δεν ακούσαμε πολλά, αλλά αυτά που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα είναι πολύ ασαφή και δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να καταλήξουμε σε κάποια ε, άποψη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της εργασίας της Europol. Είναι λυπηρό και δεν είναι η πρώτη φορά κύριε Πρόεδρε που βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης που δεν φταίει είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε ή κάποιο άλλο θεσμικό όργανο ή κάποια άλλη υπηρεσία και οργανισμό στην Ευρώπη, αλλά εμείς, εμείς ε, δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες τις οποίες χρειαζόμαστε και για τις οποίες, τις οποίες δικαιούμαστε. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω, γιατί θα πρέπει οι συμφωνίες, οι ρήτρε και τα κριτήρια τα οποία έχουν αποφασίσει για την διασφάλιση των ε, δεδομένων που αφορούν τους πολίτες μας διασφαλίζονται και θέλουμε και κάποιες απαντήσεις από τους εκπροσώπους μας. E Κύριο Σταβάρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την ε, κοινή εποπτική αρχή και την κυρία Κρούθ ιδιαίτερα για την παρουσίαση της έκθεσής της. Καταρχάς πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ολόκληρη την έκθεση συμπεριλαμβανομένων και των ε, τμήματων των μερών που είναι εμπιστευτικές, οι απόρριτες. Ε, πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε ολόκληρη την έκθεση. Ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια καινούρια μάχη, μάλλον θα σημαίνει αυτό, προς το Συμβούλιο για να έχουμε πλήρη πρόσβαση σε αυτή την τεκμηρίωση. Αφενός μάχη μέσα του Συμβουλίου και αφετέρου η εποπτική αρχή ε, στην Ουάσιγκτον, όπου θα πρέπει να πάει κάποιος να ερευνήσει το θέμα επιτόπου, να δει τι κάνουν οι Αμερικανοί. με μεγάλη δυσκολία ζητήσαμε το όνομα αυτού του ανθρώπου που είναι ο σύνδεσμος και με μεγάλη δυσκολία να αποκαλυφθεί το όνομα του ανθρώπου αυτού, του υπεύθυνου αυτού, του εκπροσώπου. Αυτός ο εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί πρέπει το όνομα αυτού του συνδέσμου να τηρείται μυστικό δεν καταλάβαμε και είχαμε και μεγάλη δυσκολία να το ανακαλύψουμε πρέπει να κάνουμε μία συνεδρία διακλεισμένων των θύρων και να καλέσουμε αυτό το άτομο να, μας, να έρθει να μας εξηγήσει, να μας ενημερώσει τι γίνεται. Από πλευρά, τώρα μέσα στην έκθεση υπάρχουν καινούργια στοιχεία για τα οποία θα πρέπει να ενημερωθούμε. Άρα λοιπόν κακός ιονός για τις μελλοντικέ εξελίξεις σε αυτό τον τομέα. Δεν νομίζω τα πράγματα πάνε καλά. Εδώ ε, υπάρχει το στοιχείο της εμπιστοσύνης. Ε, το κοινοβούλιο είναι ένα σώμα και έδειξε την εμπιστοσύνη του την συνεργασία με τους εταίρους τους όταν έγιναν οι διαβουλεύσεις ε, για τη συμφωνία SWIFT, οι διαπραγματεύσει για τη συμφωνία SWIFT είναι θέμα εμπιστοσύνη. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε γρήγορα. Ελπίζω η Κομισιόν και το Συμβούλιο να σημειώσουν αυτέ τι παρατηρήσει. Πρέπει επίση να δούμε τι γίνεται με την εφαρμογή τη συμφωνία SWIFT, ότι ενδέχεται να υπάρξει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή προσφυγή σε κάποιο εθνικό δικαστήριο. Τώρα επί του περιεχομένου, όπως μας το παρουσίασε η κυρία Κρούθ, το πιο ανήσυχο στοιχείο που μας είπε είναι ότι εκκρεμούν ήδη 8 αιτήσει. Ε, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε ήδη 8 φακέλους, 8 αιτήσει, 8 αιτήματα ε, ε, και μέσα στο πλαίσιο αυτού του προβλήματος για τη μαζική διαβίβαση στοιχείων, οι Αμερικανοί πάντα λέγανε ότι τα χρειάζονται αυτά οπωσδήποτε. Ε, τι θα γίνει λοιπόν με αυτούς τους φακέλους τώρα. Αυτά τα ντοσιέ καλύπτουν ένα χρονικό διάστημα, τα δεδομένα που είναι μέσα στους φακέλους αυτούς καλύπτουν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ορισμένες συγκεκριμένες περιφέρειες, επικράτειες και πιστεύω ότι δεν, είναι, δεν υπάρχει σωστή αναλογικότητα. Υπάρχει μια ανισορροπία ε, των σχέσεων σε αυτό το τομέα που πιστεύω ότι μπορεί να καταλήξει σε προσφυγή στα δικαστήρια. Τώρα όσον αφορά αυτά που ακούσαμε για προφορικές συμφωνίες, Καμία προφορική συμφωνία δεν μπορεί να υποπτευθεί ούτε από το Κοινοβούλιο ούτε από καμία άλλη αρχή, εποπτική αρχή, θεσμική αρχή. Ε, δεν υπάρχουν λοιπόν πρακτικά μεταξύ αξιωματούχων που συζητούν θέματα ασφάλειας. Δεν υπάρχουν πρακτικά, άρα δεν είναι υπόλογοι λοιπόν ε, οι αξιωματούχοι αυτοί στους πολίτες μας. Και Υπάρχει επίσης και το θέμα της άρνησης, της διάψευσης από πλευράς Αμερικανών ότι π.χ. αυτά ουδέποτε ελέγχθησαν. Ε, γι' αυτό λοιπόν όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι έχουμε ε, τρία πράγματα, τρεις ασυμφωνίες, τρία πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν μεταξύ αυτά που λέει η έκθεση και αυτά που συμβαίνουν τώρα επίσης ε, ότι δεν υπάρχει αίτηση των Αμερικανών να γίνουν ε, έλεγχοι και ε, εποπτείες, να γίνει μια, εποπτική, μια επιθεώρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα στοιχεία, τα στοιχεία. Δεδομένα όταν λέμε μαζική ε, μαζικά δεδομένα. Τι εννοούμε, 5-10 χιλιάδες ε, ε κυκλοφορίας ε, κονδυλίων πιστώσεων χρηματοδότησης. Ποιος είναι ο όγκος αυτών των δεδομένων. Επίσης υπάρχει περίπτωση και ποια είναι τα επιχειρήματα απόρριψης ενός αιτήματος. Στο παρελθόν όταν ζητήσαμε τέτοιες πληροφορίες δεν είχαμε ξεκάθαρη απάντηση. Και τώρα από τους μία γεγραμμένους ο κύριος Μπρόνς για να κλείσουμε το γύρο των ομάδων είμαι βέβαιος ότι θα είστε σύντομος εσείς. Δεν ξέρω αν είχε την ευκαιρία η ΚΕΑ να ελέγξει τους τελευταίους έξι μήνες ε, και τέσσερις ήταν οι αιτήσει είπατε. Αλλά τι δεν καλύψατε. Κάποιες ενοχλητικές πρακτικές ε, των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα με τη συγκατάθεση της ε, Europol που είναι ακόμα χειρότερο. Πρώτον, αυτό που ε, παρουσιάζεται ως αφηρημένη φύση των ετοιμάτων. Τι θα πει αυτό, ότι ήταν μαζικά δεδομένα δηλαδή και έτσι δεν μπόρεσε ούτε η Ευρωπόλ ούτε η ΚΕΑ να εξακριβώσει αν ήταν σύνομα όλα αυτά. Μα τότε θα έπρεπε να είχατε απορρίψει το αίτημα μέχρι να βεβαιωθείτε ότι ήταν σύνομο. Και τι θα πει προφορική ενημέρωση από τις Ηνωμένε Πολιτείες προς τη Europol χωρίς τίποτα γραπτό. Ε, πώς θα τα έλεγξει αυτά η IKEA. Σε αυτή την περίπτωση η Europol θα έπρεπε να είχε αρνηθεί το αίτημα είτε να είχε αρνηθεί ε, το προφορικό της υπόθεσης και παρά ε, τα όσα ήθελαν οι Αμερικανοί να είχε κρατήσει σημειώσεις. Και τι είναι αυτό, η Europol ε, κάνει δάνειο στο εαυτό της, μάλλον έχει καταντήσει ε, κρατικός λειτουργός των ΗΠΑ. Τι φοβούνται μακροπρόθεσμα. Είναι πολύ σημαντική βεβαίως και η πρόληψη και η αποτροπή ε, τρομοκρατικών ενεργειών. Αλλά αυτό θα πυροδοτήσει κάποιες άλλες εξελίξεις και θα μειωθούν ε, οι αντιστάσεις μας και θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε όταν μας ζητάνε δεδομένα για τελείως διαφορετικό σκοπό ή χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Πριν ε, ανοίξουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων, είναι δίκαιο και σωστό να ακούσουμε τις απαντήσεις κυρίας Κρούς, διότι ακούστηκαν πολλές επικρίσεις και πολύ σημαντικότερο νομίζω είναι ότι καταλαβαίνετε και για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι επικρίσεις. Η γενική αίσθηση της Επιτροπής μας είναι μια δυσφορία και έλλειψη ικανοποίησης από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα και τον τρόπο με τον οποίο η Europol ασκεί κάποιες δραστηριότητες με τις οποίες συμφωνήσαμε. Είμαι βέβαιος ότι θα ε, μας τα πείτε αυτά μέχρι να ακούσουμε αύριο ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ε, βουλευτές ε, για τις ερωτήσεις τους. Ήθελα να πω ότι η επιθεώρηση έγινε, ο έλεγχος έγινε τον Νοέμβριο. Η ομάδα που πήρε μέρος στην επιθεώρηση αυτή ε, έκανε μια πρώτη παρουσίαση στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου και ούτως ή άλλως υπάρχουν τριμηνιές συναντήσεις. Έγινε μια έκτακτη ολομέλεια τον Ιανουάριο για να υιοθετηθεί η, έκθεση. Όπως σας είπα έπρεπε να ενημερώσουμε την Europol και να δώσουμε μια προθεσμία για να απαντήσει. Απήντησε η Europol μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, άρα την 1η Μαρτίου υιοθετήσαμε την έκθεσή μας και τη στείλαμε αμέσως στο Κοινοβούλιο. Επομένω δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση. Αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσω. Επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα για τα οποία πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Είπατε κατά πόσο, θα πρέπει να κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευόμαστε την Europol. Δεν θέλω να είμαι άδικη. Τα 13 αυτά χρόνια της κοινή εποπτικής αρχής, μάλλον εμείς θεωρούμε ότι η Europol είναι ένας από τους οργανισμούς που προστατεύει καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα. Ε, γίνονται ετήσιες ε, επιθεωρήσεις, ετήσιοι έλεγχοι, γίνονται μετά ε, περαιτέρω έλεγχοι μετά τις συστάσεις που κάνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι η Europol συμμορφώνεται, αλλά ούτως ή άλλως η Europol συμμορφώνεται με όλους τους νόμους του σχετικού με την προστασία των δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε στην, λέει στην έκθεσή του ότι η Europol πρέπει να εξακριβώνει την νομιμότητα των ετοιμάτων και το όργανο αυτό ανέκαθεν λέγαμε ότι πρέπει να είναι ένα νομικό όργανο, ένας νομικός οργανισμός και όχι η, η Europol. Εδώ έχουμε μπλέξει λίγο τους ρόλους. Η Europol ε, πρέπει να έχει σχέσεις ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείες για να μπορεί να δέχεται και να δίνει δεδομένα ε, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Βέβαια, τα πράγματα έχουν μπερδευτεί λιγάκι, είναι κάπως συγκεχημένη η κατάσταση. Η Europol θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια επιβίωσής της μέσα σε αυτό το κάπως μπερδεμένο περιβάλλον. πρέπει να υπάρχει ένα, μια, ένας οργανισμός, μια υπηρεσία εποπτική η οποία θα ελέγχει την ε, προστασία των δεδομένων. Τώρα το πρόβλημα όσον αφορά την νομιμότητα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λύσει ε, μια άλλη αρχή, μια νομική αρχή τέλος πάντων. η Europol είχε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα για να μπορέσει να απαντήσει στις ε, απαιτήσεις και στα αιτήματα μάλλον για την ανταλλαγή των δεδομένων. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι διατάξεις της ε, συμφωνίας είναι αρκετά ε, περίπλοκες και το πρόβλημα ήταν ότι η Κομισιόν αρνήθηκε να ερμηνεύσει τις διατάξεις. Και αυτό είναι πρόβλημα γενικότερο, διότι προφανώς τελικά καταλήξαμε στο να μην έχουμε δεσμευτικούς κανόνες ερμηνείας. Τώρα, όσον αφορά την εμπιστοσύνη στη Europol, ε, χτες χτες ε, στείλαμε τις συστάσεις μας και πρέπει να σας πω ότι η Europol στην απάντηση που έδωσε δεν αρνείται αυτά τα οποία είπαμε και στην απάντηση του διευθυντή της Europol ο διευθυντής μας λέει ότι υιοθετήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις συστάσεις μας. Και σε ένα σημείο λέει, και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, ότι από τα 8 αιτήματα τα οποία υποβλήθηκαν, τα 5 αφορούσαν, που αφορούσαν στις ΗΠΑ έπρεπε να ελεγχθούν όσον αφορά την νομιμότητά τους. Ελέγχουμε κατά πόσον ε, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να υποβληθούν και γραπτά. Πάντως αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας, γιατί πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε τα στοιχεία αυτά. Είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι εδώ στη διάθεσή σας, δεν είναι απόρριτο. Δεν βλέπω γιατί, θα πρέπει, γιατί δεν θα πρέπει μάλλον να ανακοινοποιήσουμε την απάντηση της Europol στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και για σας να δείτε τι κάνει, τι προσπαθεί να κάνει η Europol ε, σαν απάντηση στις, στα αιτήματά μας, στις συστάσεις μας. τώρα για τις συναλλαγές, γιατί ε, προφανώς είναι εκατομμύρια αυτές. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. You want to add a point? Do it. Έχετε να προσθέσετε τίποτα άλλο, ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 11 Νοεμβρίου, όταν είχαμε πάει στη Europol, ασχολήθηκα εγώ προσωπικά και με τα διαδικαστικά, με τις μεθόδους ε, ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που είχαν από τα μέσα Ιουλίου και μέχρι την 1η Αυγούστου που ετέθησε η συμφωνία και στο μεταξύ έχουν οξυνθεί και βελτιωθεί οι διαδικασίες αλλά κατά την άποψή μου απομένουν δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι αυτό που ακούστηκε ήδη, ότι οι πληροφορίες που έρχονται από τις Ηνωμένε Πολιτείε. και ε, ε, δεν ε, είναι επαληθεύσιμες ή δεν μπορούν να επαληθεύονται 100% ούτε από την ΚΕΑ ούτε από την Europol με ξεχωριστό ε, επόπτη για τα προσωπικά δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και κατά πόσο ενεργά μπορούν να συμμετέχουν οι υπάλληλοι της ε, Αρχής Προστασίας Δεδομένων στην Europol την ίδια. Κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά ε, δεν τους ακούνε πάντα ε, εκείνοι που χειρίζονται αυτά τα θέματα, ούτε ο διευθυντής ε, της Europol. Δεν τους παίρνουν αρκετά σοβαρά υπόψη εκείνους που ασχολούνται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και είναι δύσκολος ο έλεγχος και στο εσωτερικό της Ευρωπόλ και για μας που είμαστε εποπτικό όργανο. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Μερικοί από εσά φαίνεται να πιστεύουν ότι η Europol ξέρει 100% ε, τι στοιχεία διαβιβάζονται με το SWIFT στι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν ισχύει αυτό. Ορισμένες κατηγορίες δεδομένων μπορεί να δίνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για συγκεκριμένες περιφέρειες και για μαζική διαβίβεση δεδομένων. Αλλά δεν δίνει το πράσινο φως από μόνη της η Ευρωπόλ για τη διαβίβαση των στοιχείων κατόπιν αιτήματος. Ευχαριστώ κύριε Ντομπίκελε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα σημαντικότερα ακούστηκαν ήδη πιστεύω. Ε, θα ήθελα να προσθέσω το εξή μόνο. Βέβαια, η έρευνα της ΚΕΑ ε, ε, θα πρέπει να ειδωθεί συνολικά και όχι ξεκομμένη από την αξιολόγηση της συμφωνίας TFTP. Αύριο ε, θα έχετε και την επιπλέον ενημέρωση για να έχετε την πλήρη εικόνα. Είναι ένα μόνο τμήμα ε, αυτό που συζητούμε σήμερα και είναι επικίνδυνο με βάση ένα και μόνο στοιχείο να αποφαίνεται κανείς για όλη την έρευνα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και εγώ κάτι που είπε η πρόεδρός μας. Δεν είναι ε, προφανές μια επιχειρησιακή υπηρεσία αστυνομίας να αξιολογεί ένα αίτημα. Εμείς στα δικά μας κράτη που είναι κράτη δικαίου τα έχουμε αναθέσει αυτά σε δικαστές ανεξάρτητους. Η Europol είναι αστυνομία. Ε, δεν μπορεί να επιφορτίζεται με τέτοια θέματα. Είναι ένα επιχειρησιακό όργανο. Ε, είναι πολύ δύσκολο να αξιολογεί και να ε, υποκαθιστά έναν ε, ανεξάρτητο δικαστή. Δεν μπορεί μια επιχειρησιακή αστυνομία να κάνει τέτοιες αξιολογήσεις. Θα ήθελα και αυτό να σας το πω για να το έχουμε υπόψη μας για περαιτέρω αξιολογήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα ορισμένα μέλη να μιλήσουν. Αλλά επειδή είναι μερικά τα θέματα που έχουμε ακόμα να πούμε, ε, πριν απαντήσουν ε, οι Ομιλητέ του πάνελ. Παρακαλώ κάθε βουλευτή να τηρεί το δίλεπτο. Ο κύριο Κοέγιο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, λυπάμαι που πρέπει να πω ότι είχα δίκιο. Όταν ε, έπρεπε να εξετάσω εκ μέρους του Κοινοβουλίου τις ε, αρμοδιότητες της Europol και το νέο αυτό ρόλο της ε, Europol το οποίο καταψηφίσαμε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου όταν ψηφίσαμε επί του θέματος και με αυτά που ακούω τώρα ανησυχώ ακόμα περισσότερο. Τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Καταρχάς ορισμένα έγγραφα ε, χαρακτηρίστηκαν ε, εμπιστευτικά πριν από μία εβδομάδα με απόφαση της ε, ΚΕΑ. Η κυρία Κρούς είπε ότι υπάρχουν προβλήματα και ότι θα ξεπεραστούν αργότερα. Αλλά πρέπει να ρωτήσω, έγινε κάποια προσπάθεια να περιοριστεί ο ρόλος Τη ΚΕΑ, τη κοινή εποπτική αρχή από του Αμερικανού. Όταν το ρώτησα μου είπαν όχι, καμία προσπάθεια περιορισμού του ρόλου της ΚΕΑ δεν έγινε από, από την Αμερικανική πλευρά. Τώρα ε, ορισμένα μέλη είπαν ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά. Και πολύ ανησυχητικό είναι επίσης αυτό το οποίο ελέγχθη όσον αφορά την επιχειρηματολογία για την νομιμότητα όλης αυτής της διαδικασίας. Τα επιχειρήματα βασίζονται, τα επιχειρήματα τα οποία ελέγχθησαν, ελέγχθησαν προφορικά και δεν υπάρχει καμία καταγραφή του τι ελέγχθη ούτε πρακτικά. Και είπε και η κυρία Κρούζ ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ότι δεν διαβιβάζονται στις Αμερικανικές αρχές ε, περαιτέρω ε, συμπληρωματικά δεδομένα από πλευράς Europol, το οποίο είναι καθαρή παραβίαση της συμφωνίας. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν έχει αισθανθεί καμία, κανένα πρόσκομα σε εργασίες της. Κύριος Λαπρινίδης, δύο λεπτά. Uh, uh, Είναι σαφές από αυτό που έχουμε ενώπιόν μας ότι η Europol κατά την άποψή μου δυστυχώς παραβίασε αυτά που τις είχαμε αναθέσει βάσει της συμφωνίας. Στο άρθρο 4 ορίζεται σαφώς ότι χρειάζεται η Ηνωμένε Πολιτείε να προβούν σε ένα αίτημα, αλλά θα πρέπει να το ε, κρίνει αυτό το αίτημα η Europol, αν θα δώσει συνέχεια. Το κοιτάτε, ό,τι σας επιτρέπουν να ε, δείτε. Αν θεωρείτε ότι το αίτημα είναι πολύ ε, ασαφές, η Europol κάπου θα πρέπει να το αξιολογεί αυτό και να λογοδοτεί. Θα έπρεπε εκεί να είναι το όργανο που ελέγχει. Εγώ και άλλοι πολλοί είπαμε όχι. Δεν θυμάμαι πια πόσοι μας πίεσαν τότε. Ε, ασκήθηκε μεγάλη πίεση. Ποιος ήταν ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι τονίσαμε τότε όμως ότι ήταν γελίο. Αυτοί που θα υποφελούνται από οποιαδήποτε πληροφορία ε, αξιολογήτω να ε, αποφασίζει να είναι κριτής και κρινόμενος αν θα πρέπει να διαβιβαστούν τα στοιχεία ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ που ήρθαμε τώρα, ας μην συγχαίουμε ε, κατά τα άλλα συνάδελφοι τα δύο που έχουμε. Έχουμε τη Europol που υποτίθεται ότι στην αρχή θα κρίνει αν θα πρέπει να δοθεί συνέχεια σε ένα αίτημα ε, των Αμερικανών. Εντάξει, αυτό το εξετάζει η Europol. Τι κάνει από εκεί και πέρα το Υπουργείο Οικονομικών ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και ο σύνδεσμος κοιτάει ε, ότι ε, την χάνουν του σωστού χειρισμού. Αυτά που κάνουν οι δικοί μας άνθρωποι εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που κατά τα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουν και δεν τα ξέρουμε, ε, είναι διαφορετικά. Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δεν ξέρω, οι συστάσεις που έχετε κάνει είναι πολύ ευρείε. Συγγνώμη, Πρόεδρε, τελειώνω. Ίσως θα πρέπει να είναι προφανέ ότι όλε οι ανακοινώσει, ακόμα και οι προφορικέ τη Europol, πρέπει να καταγράφονται από την ίδια τη Europol. Κάποιο να μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνο και να γράφει σε ένα ε, υπολογιστεί ότι ο α, ο β μου είπε το ένα και το άλλο. Ε, αυτά να είναι πρακτικά, να καταγράφονται και για τους δύο, και για την Europol και για μας. Να είναι διαβαθμισμένα, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα είναι προφορικά και τίποτα δεν καταγράφεται. Κατευθυντήριες γραμμές ε, και ποιος θα τις ερμηνεύει ε, της κυρίας Κρούς. Θέλω από κι άλλα, πρόεδρε, αλλά χρόνο δεν έχω. Ευχαριστώ. Η κυρία Νετβέλτ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους όσους ε, προετοίμασαν αυτή την τόσο κρίσιμη έκθεση και εσείς πραγματικά κάνετε τη δουλειά σας ε, σαν φύλακα αν θέλετε. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι το έργο σας. Ο κύριος Ράιτ όμως ε, πραγματικά δεν έκανε καλό σαν εαυτό του όταν αρνήθηκε να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν βρίσκεται αυτό στο στόχαστρο. Ε, ε, όσον αφορά τις διαδικασίες, ακούστηκαν πολλά. Εγώ θέλω να κάνω κάποιες, ε, κάποια ερωτήματα. Καταρχάς, είχατε κάποιες υποψίες κάποια στιγμή ότι εκτός από την μεταφορά των δεδομένων που γίνεται μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας υπάρχουν διμερείς μεταφορά δεδομένων από τα κράτη-μέλη στις Ηνωμένες Πολιτείες δεδομένα SWIFT. Επίσης έχουμε, έτοιμ, έχουμε πληροφορίες για τα αιτήματα της Europol τα συνηθισμένα αιτήματα της Europol προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για, τις, ε, για πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα αντίχνευσης της χρηματοδότηση τη τρομοκρατίας, δηλαδή για έρευνες που γίνονται στην Ευρώπη. Γιατί ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω ε, και δεν είμαι ειδικό βέβαια, είναι ότι εάν ε, υποβάλλονται αιτήματα κάθε μήνα, με κάποια περιοδικότητα δηλαδή, Πώς δεν το δικολογούμε αυτό. Δηλαδή οι τρομοκράτες είναι τόσο τακτικοί που στις αρχές του μήνα ας πούμε οργανώνουν τις δραστηριότητε τους. Ε, δηλαδή αν υποβάλλονται αυτά τα αιτήματα με περιοδικότητα δεν είναι ε, συγκυριακά, είναι κάτι το οποίο είναι, γίνεται με, με τακτικό ρυθμό δηλαδή. Επίσης, εμείς έχουμε εμπιστευτεί τις, τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όχι με τόσο, τόσο ένθερμα. Αλλά έχω την, εμπιστοσύνη, την ε, εντύπωση ότι αυτή η εμπιστοσύνη ε, δεν εκτιμάται με τον τρόπο που θα έπρεπε από τα άλλα θεσμικά όργανα. Επίσης, το συμπέρασμα στο οποίο θα πρέπει να καταλήξουμε είναι ότι επιγόντως χρειαζόμαστε μια, μια πρόταση από την ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, εξαγωγή, αν θέλετε, των δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πρόταση πρέπει να βγει σήμερα, αύριο τέλος πάντων. Επίσης, ένας γερουσιαστής, ένας βουλευτής των Ηνωμένων Πολιτειών πρότεινε μια πάρα πολύ σοβαρή ποινή, σοβαρή ποινή για αυτούς που καταχρώνονται των προσωπικών Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να υιοθετήσουμε και στην Ευρώπη. Η κυρία Έρνστ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ας πούμε ότι τα δεδομένα έχουν μπει στο μαύρο κουτί και όλες αυτές οι ανησυχίες, οι φόβοι που είχαμε στο παρελθόν για την Ευρωπόλ έχουν επιβεβαιωθεί, όλα αυτά τα έχουμε πει και τις επιφυλάξεις μας τις έχουμε εκφράσει. Ε, ε, Υποστηρίζει, υπογραμμίζω αυτά που είπατε κυρία Κρούς για τη θέση της Ευρωπόλ και αυτό το συγκεχημένο ρόλο και ή δυνατόν μια δικαστική διευθέτηση. Όσον αφορά τώρα τη μόνιμη αυτή ομάδα προστασίας δεδομένων που είπατε που θα εξετάσει τα αιτήματα από αμερικανικής πλευράς, ωραία και καλά, αλλά αυτό που δεν μας είπατε είναι αν αυτή η ομάδα που συστάθηκε ε, έλαβε θέση υπέρ ή κατά αυτό των ετοιμάτων Δηλαδή ποιο ήταν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της εργασίας αυτής της ομάδας την οποία συνθέσατε. Αυτό δεν τα ακούσαμε. Και επίσης είπατε ότι εξέτασαν 8 αιτήματα, 8 και τα πέντε αφορούσαν στη, ε, παροχή συμπληρωματικών δεδομένων, οι άλλοι τρεις φάκελοι τι έτοιμα είχαν, περίχαν. Ο πρόεδρος η κυρία Αργεντίνη, Αρχεντίνη, συγγνώμη, σας ξέχασα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω πολλές ε, κριτικές ερωτήσεις για τη Europol και αν έχουν τηρήσει τις συμφωνίες ή όχι. Πρέπει να τεθούν αυτές οι ερωτήσεις, αλλά εμείς να αναρωτηθούμε. Πριν το καλοκαίρι το Κοινοβούλιο συμφώνησε χωρίς τους πρασίνους να στέλνει μαζικά δεδομένα από ευρωπαϊκούς τραπεζικούς λογαριασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπαμε, αυτό ήταν η πρόφαση, ότι θα στείλουμε και κάποιον στην Ουάσιγκτον να τα ελέγχει αυτά. Και το ξέραμε ότι η Europol δεν θα ήταν σε θέση να τα ελέγχει όλα αυτά. Το ξέραμε από τότε. Και μας είπανε ε, και τι αξιολόγηση και τι παρακολούθηση θα γίνεται, γραπτή, προφορική κτλ. Συμφωνώ και εγώ ότι δεν γίνεται ε, αυτά να γίνουν προφορικά. Παρόλα αυτά, παρόλο που ξέραμε ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει, τα δεχτήκαμε. Και τώρα η Europol θα τηρήσει το άρθρο 4 της συμφωνίας ή όχι. Δεν έχει έρθει η ώρα να συνέλθουμε και να πούμε ότι δεν στέλνουμε μαζικά δεδομένα των πολιτών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα πολιτών που δεν έχουν κάνει τίποτα κακό, τίποτα επιλήψιμο. Θέλω να ευχαριστήσω την κοινή εποπτική αρχή για την ενημέρωση, αλλά ε, το πρόβλημα, το έλλειμμα είναι δικό μας. Ευχαριστώ. Κυρία Σίπελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές επικρίσεις ακούστηκαν Γι' αυτό θα περιοριστώ σε, ορισμένες, σε λίγες ερωτήσεις και ορισμένες υποδείξεις. Οι πληροφορίες που μας έδωσαν δεν είναι συγκεχημένες. Γι' αυτό πρέπει να ξαναρωτήσω. Το SWIFT κάνει επεξεργασία των δεδομένων τα εκατομμύρια των δεδομένων που λαμβάνονται προέρχονται από εκατομμύρια πολίτες ή προέρχονται από μαζικούς οργανισμούς, φορείς, ε, εταιρείες ή οποιαδήποτε άλλη αρχή. Ο SWIFT δεν μπορεί να εξετάσει την, τις κατηγορίες στις οποίες υπόκεινται τα δεδομένα. Γι' αυτό είναι σημαντικό η αμερικανική πλευρά να μας απαντήσει καταρχάς πώς διαχειρίζεται ε, τα δεδομένα και η Ευρωπόλ να εξετάσει εμπεριστατωμένα εάν υπάρχουν αιτήματα τα οποία δικαιολογούν ε, μια τέτοια ερώτηση. Η Ευρωπόλ οι πληροφορίες ε, δεδομένα αυτά είναι πολύ σημαντικά και για τον εκπρόσωπο, και τον υπεύθυνο, ο οποίος κάθεται στο Υπουργείο Οικονομικών και εξετάζει αυτά τα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε ε, τι ακριβώς δεδομένα, με ποια δεδομένα ε, δικαιολογείται η έγκριση του φακέλου, η έγκριση του αιτήματο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε τι προσόντα θα έχει ο, ο υπεύθυνος, ο αρμόδιος για τη διαχείριση αυτών των δεδομένων και την εξέταση των φακέλων στο Αμερικανικό Υπουργείο τι προσόντα πρέπει να έχει, θα είναι τεχνοκράτης, θα είναι ειδικό ε, για, τα δεδομένα, στα ηλεκτρονικά, σε τι. Τελευταία κυρία Λάτφορτ και μετά απαντήσεις. Thank you, Chairman. I hope last but not least. Ευχαριστώ, Πρόεδρε είμαι τελευταία που έχω το λόγο. Εγώ νομίζω ότι είχαμε δίκιο να υπερψηφίσουμε τη συμφωνία υπό το φως των ρητρών ασφαλείας τις οποίες είχαμε προβλέψει, είχαμε ζητήσει, αλλά νομίζω μας πρόδωσαν. Εγώ εκφράζω μια διαφορετική πλευρά από τον κύριο Λαμπρινίδη και πιστεύω όταν εξετάσαμε το θέμα αυτό πέρσι, τα φαινόμενα ήταν, ήταν ξεκάθαρα ότι θα ξεφύγει ότι θα προδοθούμε, ότι θα μας ξεφύγει από τα χέρια μας. Ε, δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Αυτό το επιβεβαιώνει η έκθεση, η οποία όμως σοκάρει, ακόμα περισσότερο, μας σοκάρει διότι προδίδει, μάλλον ε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει πια εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ πιστεύω ότι βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, ανταλλαγή δεδομένων για θέματα τρομοκρατία, αλλά πρέπει να είναι αξιόπιστες οι ρήτρε ασφαλείας τι οποίε ζητήσαμε. Ρήτρες ασφαλείας, αυτές πρέπει να είναι 100% αξιόπιστες. Όσον αφορά τώρα αυτό το μυστικό παράρτημα, το απόλυτο παράρτημα, τι είναι αυτή η διαδικασία. Η Ευρωπόλ χαρακτηρίζει ω απόρριτα παραρτήματα τα οποία οποία αναφέρονται στο μηχανισμό της Europol για την εφαρμογή του άρθρου 4. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να, το δεχτούμε αυτό. Η Europol να χαρακτηρίζει απόρριτες δικές της διαδικασίες. Ε, είναι πολύ απογοητευτική αυτή η έκθεση γιατί δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε. Όσον αφορά τις διάφορες συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων. Για αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν, από το Συμβουλίο, το Υπουργείο Οικονομικών. Θα ήθελα μάλλον να έχω εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους φορείς, να υπερισχύει η εμπιστοσύνη, αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα η θέση μας δυσκολεύεται ε, ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Τώρα φτάσαμε στα συμπεράσματα και θα ακούσουμε τον τελευταίο λόγο από την κυρία Κρούθ, και είμαι βέβαιη ότι θα αναφέρετε όλα αυτά τα οποία ελέγξησαν στον κύριο Wainwright ε, στο διευθυντή της Europol και να το μεταβιβάσετε αυτές τις ανησυχίες, τις επιφυλάξης που, που ακούστηκαν εδώ όσον αφορά την έξεση. Ελπίζω, θα έχουμε βεβαίω τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα αυτό και με την αρμόδια επίτροπο Κυρία Ιντεβέλτ, διαδικαστικό, τι, τι θέλετε. Πολύ σύντομα, ο κύριος Βένρετ θα πρέπει να ξανάρθει στην Επιτροπή μας. Να τον προσκαλέσουμε να ξανάρθει, διότι υπάρχουν ερωτήματα τα οποία μόνο αυτός μπορεί να απαντήσει. Ο πρόεδρος, ε, ναι, ναι, πιστεύω ότι αυτό είναι κοινό αίτημα. Ε, έτσι πιστεύω και εγώ. Όσο νωρί, νωρί ταχύτερα, τόσο καλύτερα να προσκαλέσουμε και πάλι τη θητή της Europol. Κυρία Κρούθ, για να, για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε για να απαντήσω τώρα στον τελευταίο γύρο των ερωτήσεων. Μία ερώτηση αφορά άλλες, τυχόν άλλες διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών ε, και αμερικανικής πλευράς ε, όσον αφορά τις ε, μεταφορά χρημάτων ή χρηματοδοτικέ ε, συναλλαγές. Έχουμε με άλλε διμερεί συμφωνίε αλλά αφορούν τον τουρισμό. Δύο. Δύο. Δύο συμφωνίε τώρα υπογράφτηκαν ή θα υπογραφούν ε, σύντομα από κράτη-μέλη που αφορά το, το προφίλ των τρομοκρατών, ανάλυση προφίλ τρομοκρατών και επίσης ζητήσαμε μία Ευρωπαϊκή Συμφωνία ε, για το θέμα αυτό και δεν ξέρω αν θα το ολοκληρώσουμε. Τώρα, ε, η αρχή μας εξέτασε το άρθρο, το άρθρο 10 του TFTP ε, και η Europol έχει εντολή να εξετάσει τα άρθρα 9 και 10, εάν τα άρθρα 9 και 10 της συμφωνίας τηρούνται, γίνονται σεβαστά. Λοιπόν, είναι και αυτό έργο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας TFTP. Και αυτό θα το στείλουμε, θα στείλουμε αυτό το αίτημα ε, όσον αφορά το δημοσιευμένο, το δημόσιο μέρος της έξεσης. Το μη διαβαθμισμένο ε, για το θέμα του αρμόδιου για τα δεδομένα. Η Europol έχει 48 ώρες καταγραφής των δεδομένων και ξέρουμε ότι ε, δεν τηρούνται πάντοτε τα στάνταρ αυτά τα οποία ζητάμε, μα δεν είναι και υποχρεωτικά. Η απάντηση του διευθυντού της Europol ε, στις ε, σε αυτά που του ζήτησα μου απάντησε ότι θέλει να δημιουργήσει ένα μηχανισμό όπου θα καθορίζεται γραπτός ε, η διαδικασία διαχείρισης των δεδομένων, ότι όλα αυτά θα καθορίζονται γραπτά έτσι όταν η αρχή εξετάζει και επιθεωρεί να μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα και τη θέση του αρμόδιου στο Αμερικανικό Υπουργείο. Υπάρχει κάτι το οποίο ξέχασα. Θέλω κάτι άλλο να προσθέσω. Οι αρμοδιότητες που δόθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ελέγχει τη Europol. Στις ελεγκτικές αρμοδιότητες λοιπόν. Είναι αρκετά πρόσφατες αυτές οι ελεγκτικές αρμοδιότητες επί της Europol θα δημιουργηθεί ένα κοινοβουλευτικό φόρουμ, διακοινοβουλευτικό φόρουμ με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων όπως θα συζητηθούν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και θα γίνει και ενημέρωση βεβαίως για το πώς λειτουργεί η Ευρωπόλ. Αυτό το φόρουμ θα λειτουργεί ο σύνδεσμος με όλα τα εθνικά κοινοβούλια και θα είναι δυνατόν να υπάρχει άμεση επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό θα είναι το διακοινοβουλευτικό ε, φόρουμ μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι. Διαδικαστικό, κύριο Λαπρινίδη. Σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και πάλι, κυρία Κρούζ. Εγώ έχω πρόβλημα, όχι με εσά κατά ανάγκη, αλλά και πάλι αναφέρετε κάποια έγγραφα που, δεν, που θα μπορούσατε να μας δώσετε για το τι βρήκατε, για το πώς ε, ε, χρησιμοποιεί το άρθρο 10 η Europol για τα αιτήματα. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε εκατό φορέ και χίλιε φορέ να κάνουμε την ίδια συζήτηση. Ήρθε ο κύριο Γουέν Ράιτ πριν από μερικέ εβδομάδε. Δεν μα έδωσε καμία ενημέρωση από αυτή που ήξερε προφανώ και ήξερε και η ΚΕΑ. Μα έδωσε μερικά έγγραφα από ό,τι που θυμάμαι τι ήταν κάτι άσχετα. Τώρα έχουμε άλλο έγγραφο και διαπιστώνουμε ότι αργότερα μπορεί να μα στείλουν κι άλλα. Εγώ δεν μπορώ να δουλεύω έτσι θα παρακαλούσα να έχουμε όλα τα στοιχεία όταν συζητάμε, ό,τι έχει και θα μας ε, χρειαστεί. Εν πάση να έχουμε ένα σύνολο όσο γίνεται ε, ε, συνεκτικότερο. Και τέλος, εγώ δεν ξέρω ποιος σε αυτό το κανόνα για τις 48 ώρες, Για δεν ήταν στη συμφωνία TFTP, μπορεί να ήταν και να το έχω ξεχάσει. 48 ώρες σας δίνουνε, το λέει, γιατί 48 ώρες, ορίστε, το συντομότερο λέει, ωραία, 48 ώρες έχει νόημα όταν είναι μια σούπερ κατεπίγουσα κατάσταση. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν είναι πια και η τρομερή επίγουσα ανάγκη. Και όταν μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα και θέλουμε να είναι ε, πολύ συγκεκριμένο το αίτημα, ε, τεκμηριωμένο και περιορισμένο, ε, το θεωρώ παράδεκτο να έχει δεχτεί 48 ώρες η Europol, αν τι έχει δεχτεί τις δέχτηκε και μετά να κλαίγεται ότι δεν τη φτάνει ε, το διάστημα αυτό για να δουλέψει. Αφού έχει περιοριστεί η ίδια. Μάλιστα, τα έχουν σημειώσει αυτά, όχι μόνο τις ανησυχίες που εκφράσατε, αλλά και τα προβλήματα που εκθέσατε ε, και τα προβλήματα που έχουμε εμείς και η Επιτροπή μας για να ελέγχουμε την εφαρμογή των όρων που συμφωνήσαμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε για το TFTP. Έτσι, αμέσως απευθύνουμε και νέα πρόσκληση στον κύριο Wainwright, διευθυντή της Europol, να ξανάρθει για να ξανασυζητήσουμε ακριβώς τα ίδια θέματα. Και αύριο παρουσία της κυρίας Σεσίλια Μάλμστρομ ε, της Επιτρόπου. Ευχαριστούμε όλους τους προσκεκλημένους μας που ήρθαν σήμερα. Χαίρετε και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Yes. Yes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 will be right in proceeding right away. Μάλιστα. Προχωρούμε αμέσως στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, που είναι και πάλι ένα σημαντικό ζήτημα και είναι το υπαριθμό 6. Ευρωπαϊκή Εντολή Ερεύνας ε, σε ποινικέ υποθέσεις. Έχουμε τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων και τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Very interesting dossier. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Ε, ο εισηγητής είναι ο συνάδελφος κύριος Νούνο Μέλο για την πρόταση οδηγίας για την ε, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερεύνης για ποινικέ υποθέσεις κατόπιν πρωτοβουλίας 7 κρατών μελών. Αυτή η πρωτοβουλία ε, χρειάζεται και προβλέπει μια αναγνώριση σχεδόν όλων των ερευνητικών μέτρων. Έγινε μια πρώτη συζήτηση το Δεκέμβριο όταν ήρθε ο πρόεδρος, ε, το τότε ο Βέλγος Υπουργός Δεκλέρκ και μας παρουσίασε αυτή την πρόταση. Ε, χρειάζεται για αυτή την υπόθεση ε, μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Και μετά από αίτημα του κυρίου Αλβάρο, το οποίο η Επιτροπή μας εδέχτηκε, ζητήσαμε γνωμοδότηση από τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Θεμελιδών Δικαιωμάτων, τη λάβαμε, τη διανύμαμε και τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο ε, του οργανισμού, τον κύριο Γιώνας Γκρίμχεντεν, τον οποίο καλωσορίζουμε και θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του και μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή κύριο Μέλο και άλλα μέλη της Επιτροπής. Είπα ότι καλύτερα να μιλήσει πρώτα ο εισηγητής κύριος Μέλλο και μετά από την υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο κύριος Μέλλο, εσείς είστε ο πρόεδρος και έτσι αποφασίζετε, εντάξει. Μπορώ να αρχίσω. Α, θα μιλήσω πορτογαλικά. Καταρχάς, Δεν, έχω, δεν έχουμε ακόμα ε, την τελική μας ε, θέση, επίσημη θέση, λάβει για το σχέδιο έκθεσης, ε, διότι μόλις λάβαμε πληροφορίες, σημαντικές πληροφορίες για μια πρόταση κανονισμού, πρόταση Οδηγία η οποία θα έχει πολλές επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις και θα πρέπει να το σκεφτούμε σημαντικά. Ε, αυτή τη στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις. Ε, δεν θέλω να προκαταλάβω τους ομιλητές που θα μιλήσουν μετά από μένα. Θα περιμένω να ακούσω τις απόψεις τους. Θέλω όμως να τονίσω ότι αυτή η πρόταση οδηγίας η οποία έχει την υπογραφή της Επιτρόπου, κυρία Ρέντινγκ, αυτή η πρόταση επιβεβαιώνει την προηγούμενη έκθεση η οποία ήδη έχει υποβληθεί το Σεπτέμβριο αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τι θα μας πει η υπηρεσία, η αρμόδια υπηρεσία για τις θεμελιώδη δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, να περιμένουμε τη γνωμοδότησή της για να διαμορφώσουμε και εμείς την άποψή μας. Υπάρχουν από πλευράς ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Εκτελεστική ορισμένα βασικά ζητήματα. Η Κομισιόν πιστεύει ότι αυτό το μέσον ε, καλύπτει την αμοιβαία αναγνώριση των κοινών ερευνητικών διαδικασιών και λέει ε, ε, ότι, αστυνομικά μέτρα δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Πιστεύει η Κομισιόν ότι θα πρέπει τελικά να γίνει κανονισμός και όχι οδηγία. Η Κομισιόν πιστεύει ότι χρειάζεται μια ειδική αναφορά για την προστασία δεδομένων ότι οι πόροι θα πρέπει να αναφέρονται πιο λεπτομερώς, ότι το ποινικό ε, δίκαιο βεβαίως ε, έγκυται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Εδώ έχουμε ακόμα αρκετά να αποσαφηνίσουμε. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε ένα υλικό στα χέρια μας πάρα πολύ ευαίσθητο και ότι δεν υπάρχει ακόμα συνένεση επί του θέματος. Εγώ ως πρέπει να πω ότι ο στόχος μου είναι να συζητήσω με όλους τους σκιώδεις συζητητές, αν είναι δυνατόν μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα. Θα αξιολογήσουμε όλη την τεκμηρίωση και την θέση της υπηρεσίας, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Η υπηρεσία αυτή ε, προβάλλει παρουσιάζει προτάσεις και από ρεαλιστική άποψη θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σεμελιωδών Δικαιωμάτων να μας εξηγήσει κατά πόσον αυτή η νέα ευρωπαϊκή λογική ενδέχεται να βρεθεί σε αντιπαράθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή με τις διάφορες ε, με τα διαφορετικά ποινικά δίκαια τα οποία ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι από κράτο μέλο σε κράτο μέλο υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι χειρισμού ποινικών υποθέσεων. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα συναντηθώ, σα είπα, πρόθεσή μου είναι την ερχόμενη εβδομάδα με τους κοιόδη εισηγητής. Ελπίζω να υπάρχει μια κοινή βάση κατανόησης και εργασίας ε, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ενιαία κοινή θέση στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Τώρα θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανθρωπίνων ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ε, στείλω και ένα χαιρετισμό από την ε, Βιέννη. Ε, θα πω την άποψή μας όσον αφορά την τη γνωμοδότηση και μετά θα ακούσω τις απόψεις σας. Ούτως ή άλλως πολλές φορές διασυνοριακές ε, ρυθμίσεις χρειάζονται για να ε, ελέγξουμε την, ε, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχουν όμως και κάποιες ασυμβατότητες ανάμεσα στις νομικές διαδικασίες των κρατών μελών που κινδυνεύουν να παραβιάσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα μας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσουμε μια γνωμοδότηση. Ε, τον Γενάρη υπευλήθη επίσημα το αίτημα, την ε, υποβάλαμε τη γνωμοδότηση το Φεβρουάριο, 15 σελίδες, 5 κεφάλαια όπου καλύπτουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα Ε, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή έρευνα, Έρευνας ε, για την ε, δίκαια δίκη, για την προστασία των δεδομένων, για την προστασία των δικαιωμάτων. Απαντήσαμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία τέθησαν για το κατά πόσον χρειάζεται μια αναθεώρηση από πλευράς του εκτελούντος κράτος. Εδώ αναφέρουμε την ανάγκη ε, για να, υπάρχει, να υπάρχουν τα επιχειρήματα απόρριψης ε, με βάση την, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα αναφερόμαστε σε, συγκεκριμένα, ε, σε συγκεκριμένες παραβιάσεις ε, είναι, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Είπαμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία, ιεράρχηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή δεν θα αναφέρουμε κάποια θεμελιώδη δικαιώματα και θα, θα αγνοήσουμε κάποια άλλα, σαν όπως έγινε και στο σχέδιο το οποίο πήραμε. Επίσης προτείνουμε κάποιες ρήτρε διασφάλισης έτσι ώστε να ενισχύσουμε την πρόταση. Λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε τα λιγότερο διεισδυτικά μέτρα όταν αναφερόμαστε ε, στην νομική σαφήνεια. Ε, μιλάμε για την ποιότητα των διασυνοριακών ε, εντολών και οργάνων μιλάμε για την υποχρεωτική επικύρωση που θα γίνεται από κάποιον δικαστή ή εκπρόσωπο της δικαστικής εξουσίας. Επίσης, ε, ε, λέμε ότι θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση με βάση τα αποδεκτικά στοιχεία. Ε, δεν θα, το, θα αφήσουμε ας πούμε ε, ανοιχτή την περίοδο ας πούμε μια περίοδο πέντε ετών και να δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λέμε ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από την αρχή. Εάν το εργαλείο αυτό δεν ε, αποδίδει, εάν η νομοθεσία δεν αποδίδει, τότε οι συνέπειες θα πρέπει να φανούν αμέσως. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη γιατί ε, θα στηριζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα και με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει αν θέλετε μια τροχοπέδη σε επίγουσες περιπτώσεις. Επίσης ε, λέμε ότι αυτή η αξιολόγηση των συμβα... της συμβατότητας των νομικών διαδικασιών ε, θα ελέγχει τις πρακτικές που εφαρμόζονται για να δούμε και όχι μόνο τις παραβιάσεις αλλά και την, και αντίθετα και το πόσο ενισχύονται σε κάποιες περιπτώσεις τα ενισχύεται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι το 15 σέλιδο έγγραφο το οποίο υποβάλαμε. Ελπίζω να απαντήσαμε στα ερωτήματα του κύριου Μέλο προσπαθήσαμε να αντισταθμίσουμε τα πλεονεκτήματα μιας ενός διασυνοριακού εργαλείου, το οποίο θα ενισχύσει την δικαιοσύνη και που θα εξασφαλίσει ε, από τα δικαστήρια τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ελπίζουμε ότι η γνωμοδότησή μας ε, θα προσφέρει μια προστιθέμενη αξία, ε, γιατί στηρίζεται στην αντικειμενικότητά μας, στην αξιοπιστία μας, Επίσης υπάρχουν και κάποιες εκθέσεις μας, τις οποίες έχω φέρει, ε, που νομίζω ότι μπορούν να ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διεφήμιση λέει ο Πρόεδρος. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριε Άλμπρεχτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση και του εισηγητή κιόλα. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, πάρα, ήταν πιο εύκολο να ελέγξουμε τη διασυνοριακή εναρμόνιση όταν μιλάμε για καταπολέμηση του εγκλήματος ή την αλλά όταν μιλάμε όμως για εναρμόνιση θεμελιωδών δικαιωμάτων ή για την εναρμόνιση κάποιων νομοθετικών διατάξεων, εκεί τα πράγματα είναι λιγότερο εύκολα. Τώρα όμως είναι προφανές, μια και, όταν, και έχουμε και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ότι υπάρχει κοινοτική αρμοδιότητα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εμείς σαν πράσινοι θέλουμε να έχουμε ένα εργαλείο το οποίο να μας επιτρέπει την συλλογή των στοιχείων διασυνοριακά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρξει μια συνεργασία διασυνοριακή για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είδαμε ότι εκεί υπάρχει κάποια έλλειψη εμπιστοσύνης, μια καχυποψία ανάμεσα στα, στους πολίτες για τα μέτρα αυτά και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι σημαντικό όχι να μην, γίνουν οι δικαστές μηχανές συνεργασίες, συνεργασίες ε, και να υιοθετούν διαδικασίες που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε. Θα πρέπει να ε, συνεργαστούμε περισσότερο, να υιοθετήσουμε κοινούς κανόνες. Γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην καλύτερη συνεργασία και στην καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις δικαστικές ε, ε, αρχές, να, υπάρχουν άμεσες επαφέ, να υπάρχει άμεση επαφή και επικοινωνία ανάμεσα στις δικαστικές αρχές, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομοιομορφία σε αυτό το εργαλείο και να είμαστε σίγουροι ότι οι διατάξεις εφαρμόζονται σωστά και το η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα δεν θα πρέπει να διέπεται από μια οδηγία αλλά από έναν κανονισμό. Και θα ήθελα να ζητήσω στον κύριο, από τον κύριο Μέλο να προτείνει έναν κανονισμό και όχι, ένα... μια... όχι μια οδηγία, διότι με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ο ένας ελάχιστος κοινό παρονομαστής που θα μας ε, οδηγήσει και σε μια αποδοχή από πλευρά των πολιτών πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια στοιχεία που να επιτρέπουν την απόρριψη, κάποια επιχειρήματα για την απόρριψη. Μιλάμε για την αναλογικότητα των ετοιμάτων, μιλάμε για την εξοδικαστική χρήση. Ε, Μιλάμε για, τις, για ποινικέ αρμοδιότητες ε, της, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, εάν τα πάντα γίνονται δεκτά από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα απόρριψης από πλευράς ενός κράτους μέλους. Κυρίως μετά την έκθεσή σας, την παρουσίασή σας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα, όταν μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα, να ε, διασφαλίσουμε μια ικανοποιητική και αξιόπιστη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά έτσι ώστε οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να έχουν μια ομοιόμορφη εφαρμογή γιατί αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε για ενημέρωση ε, τα βλέπουμε τα πράγματα από μια άλλη προοπτική, αλλά όλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας ε, στην ε, απόφασή μας για την ε, ανταλλαγή πληροφοριών. Η, Βαρόνι η Λούντφορντ. Λοιπόν, γενικά, γενικά υποστηρίζω την αμοιβαία αναγνώριση, τα μέτρα αμοιβαίας αναγνώρισης. Το πρόβλημα είναι, όπως ξέρουμε, την τελευταία δεκαετία τα διασυνοριακά μέτρα προσαγωγής ε, δεν έχουν ε, στηριχθεί στα κατάλληλα μέτρα και δεν έχουν, ε, είχαν ικανοποιητική εξέλιξη ούτε για τους προσαγόμενους, ούτε για τους κατηγορούμενους, ούτε για τους προσάγοντες. Τέλος πάντων, πρέπει μεταξύ των 27 διαφορετικών δικαστικών αρχών ε, να υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη για να επιτύχει αυτή η διαδικασία. Ε, δεν έχουμε καμία ρήτρα σε θεμελιωδών δικαιωμάτων γιατί ξέρουμε ότι όλες οι 27 χώρες θα συμμορφωθούν πλήρως με τη σύμβαση του Στρασβούργου και, και, και την ομολογία για τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτή είναι μια ιδεατή κατάσταση και δεν θα πρέπει να δεχτούμε αυτή την ε, ωραία την δήλωση της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας ότι ο καθένας θα σέβεται, κάθε μέρος, συμβαλόμενο μέρος θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα ασφαλείας σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις καταπάτησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, από ένα τρίτο μέρος. Ε, από κάποιον τρίτον. Ε, στην ε, εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, Σύλληψης, τουλάχιστον το δικό μου κόμμα, αντίθετα από τους συντηρητικούς και στη Βουλή των Λόρδων, στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης υπάρχει μια συγκεκριμένη ρήτρα που λέει ότι ένας δικαστής μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει βάση του ευρωπαϊκού εντάλματος αυτού αν υπάρχουν σαφή επιχειρήματα κλπ. κλπ. Δεν ξέρω όμως αν έχει ολοκληρωθεί μια τέτοια διαδικασία στις, στα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σκοτία, στο, της Αγγλίας για τη σκοτία δεν ξέρω αλλά σίγουρα σε ορισμένε περιπτώσεις θα έπρεπε να είχε υπάρξει άρνηση ε, πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών απαιτεί για να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση να υπάρχει μια ρήτρα ε, άρνησης, απόρριψης. Υπάρχουν υποθέσεις, πιστεύω, όπως οι σε ε, διαδικασίες, σε ποινικές προσαγωγές, επίσης ε, το, σε θέματα του διπλού... Ε, in the case of transfer of a person, that should be a person who... in να έχουμε μια τέτοια ρήτρα ασφαλείας Επίσης να μην χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί αυτοί για την ταχύτατη απέλαση. Ε, ο κύριος Κίρκοπ, πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που η Lady ε, Λάμφορντ μας θύμισε και πάλι το σημαντικό ρόλο της Βουλής των Λόρδων στο Ηνωμένο Βασίλειο Χαίρομαι που οι Λόρδοι προσέχουν ορισμένα από αυτά τα ζητήματα σε αντίθεση με το Westminster, με την Βουλή, η οποία πολλές φορές δεν δίνει τη δέουσα προσοχή με το Κοινοβούλιο, το Βρετανικό. Καταρχάς λοιπόν η διαδικασία απελήθευσης και η αναλογικότητα, αυτό βεβαίως το έχουμε πει, Καταρχάς ε, αυτή η αναγνώριση και η αυτή η έκδοση και η διαδικασία έκδοσης δημιουργεί πολλές επιφυλάξεις διότι δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι η, η εκδούσα αρχή ποια θα είναι η αρχή που θα εκδίδει αυτό, αυτή την εντολή πρέπει να υπάρχουν σαφώς ε, ρήτρε ασφάλειας έτσι ώστε όλες αυτές οι διαδικασίες εξέτασης και έκδοσης του εντάλματος να είναι ε, ε, μη προσβλητές, απρόσβλητες. Ε, και επίσης έτσι διευκολύνεται και το έργο του, του δικαστή, της δικαστικής αρχής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα κενά και έλλειψεις. Η, το στοιχείο της αναλογίας, αναλογικότητας ε, πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ε, το είδος του εγκλήματος, παραδείγματο χάρη αν απαιτείται η εξέταση DNA ή επίσης οι τυχόν κυρώσεις που επισύρει, οι επισύρει ένα ε, έγκλημα, μια, ένα ποινικό αδίκημα. Είναι λοιπόν, πρέπει να, να, να, σεβόμαστε την αρχή της αναλογικότητας και θα πρέπει ειδικά να υπάρχουν διαδικασίες προσφυγής, να υπάρχουν ρήτρες ε, ε, ασφα, εξασφάλισης της σωστής διαδικασίας και τρίτον, ποια αρχή θα διενεργεί όλη αυτή τη διαδικασία και πού θα προσφεύγουν. Κύριο κύριος ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη γνωμοδότηση, για την έκθεση. Όντως, γίνεται ένα άλμα προς τα εμπρός για την αμοιβαία αναγνώριση, ε, με εγγυήσεις όμως. Για τα θέματα αυτά της δίωξης και της έρευνας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ε, τον οργανισμό. Όταν έχουμε προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενικά ε, θα πρέπει να δοκιμαστεί αυτή η εφαρμογή και αν υπάρχει δυνατότητα άρνησης. Όταν κάποιος δεν θέλει να προχωρήσει όμως μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό ως κολλησιεργία και μπορεί να ε, ορθώσει εμπόδια σε αυτό το άλμα που σας είπα και να προφασίζεται πάντα ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι πρέπει να το ελέγχει αυτό για θεμελιώδη δικαιώματα και να μην εφαρμόζει ποτέ την εντολή. Μα πρέπει να γίνεται αυτό για να είναι τα κράτη άψογα στη συμπεριφορά τους. Εντάξει, θα χρειαστεί χρόνο, αλλά τι να κάνουμε, κρίμα. Ε, αλλά χρειάζονται χρόνο αυτά τα πράγματα. Και η ποινική δικονομία και η διαδικασία χρειάζεται το χρόνο της. Δηλαδή, θα ήθελα να τονίσω αυτό και ένα άλλο θέμα ακόμα που ε, είναι μια ανισορροπία του συστήματος. Όταν έχουμε υπόπτους, ας πούμε, και ε, διώκονται και με ένα τέτοιο ένταλμα, εντολή έρευνας. Αν θέλει κάποιος να το προσβάλλει αυτό ένα υποπτός θα πρέπει να στραφεί κατά της αρχής που εκδίδει αυτό το ένταλμα ή αυτή την εντολή έρευνα, το οποίο ο κράτος όμως μπορεί να μην είναι η χώρα του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Και τι δικαιώματα έχουν κάποιες τρίτες ε, πλευρές, τι δικαιώματα έχει η εισαγγελία και ο ίδιος ο ύποπτος. Επίσης, η πρόταση αυτή ε, είναι μια πρόταση που ε, εξυπηρετεί τις διοκτικές αρχές. Εάν θέλει όμως και ο ύποπτο κάτι να αξιοποιήσει από αυτή τη δυνατότητα, δεν το ε, λέμε στο, στην πρότασή μας. Η εισαγγελία, ό,τι διαθέτει η εισαγγελία θα πρέπει κανονικά να διαθέτει και υπεράσπιση, έτσι δεν είναι, του κατηγορουμένου και του υπόπτου κάθε φορά. Και κάτι άλλο ε, Χρειάζονται εγγύσει λοιπόν και εγώ είμαι μάλλον επικριτικό ω προ την κείμενη πρόταση. Ευχαριστώ κύριος Παπα-Νικολάου παρακαλώ. Καταρχά, συμφωνώ ότι όλοι θα πρέπει να σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα και είμαι βέβαιο ότι και ο εισηγητή μα θα τα εξετάσει όλα αυτά. Ένα παράδειγμα ακόμα να σα δώσω για αυτό το θέμα, που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου. Εδώ και μερικά χρόνια ε, στην Ευρώπη είχαμε ένα ευρωπαϊκό σκάνδαλο, έτσι, με τη γνωστή εταιρεία Siemens στη χώρα μας, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη. Η Siemens κατηγορήθηκε ότι ε, δωροδόκησε, ότι προσπάθησε ε, να δωροδοκήσει πολιτικούς για να μπορεί να ευνοείται στις συμβάσεις. member states and have με πολλά κράτη-μέλη για να έχουν τη δυνατότητα να κανονίζουν ε, με άμεσες αναθέσεις κτλ. Μέχρι τώρα έχουν περάσει χρόνια και δεν έχουμε λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις για τις έρευνες και την ανταλλαγή ε, πληροφοριών και ενημέρωσης μεταξύ των κρατών μελών για την έρευνα προκειμένου που έχει γίνει από τις ελληνικές αρχές αλλά και από άλλες ε, ευρωπαϊκές αρχές, γερμανικές και κάποιων άλλων κρατών. Εάν καταφέρουμε να αναπτύξουμε αυτό το κανονισμό ή οδηγία, δεν ξέρω ό,τι θα είναι, ό,τι προσφέρεται, εν πάση περιπτώσει, και εμπιστεύομαι τον κύριο Μέλο που ξέρω ότι έχει πολύ μεγάλη πείρα στη χώρα του σε τέτοια θέματα, θα είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα ακριβώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το προσεχές μέλλον για να είμαστε σε θέση ε, και σε επίπεδο δικαιοδοσίας πλέον ε, να ελέγχουμε τέτοια θέματα και να έχουμε και απαντήσεις να δίνουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοτσέτα. Ε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους της νομοδότησης, διότι μας επιτρέπει να έχουμε ένα πληρέστερο πλαίσιο πληροφοριών. Και εγώ πιστεύω ότι μια Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας θα βελτίωνε τις, ε, τις δυνατότητες συνεργασίας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Όμως θεωρώ ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει σε ένα πλαίσιο βεβαιότητας. Ο μηχανισμός ο οποίος προτείνεται παραβιάζει τα, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, κατά τα μου τουλάχιστον, ε, διότι παραβιάζει κάποια εθνικά συντάγματα που δεν επιτρέπουν, παραδείγματο χάρη, οι έρευνες να γίνονται χωρίς την δικαστική άδεια. Παραδείγματο χάρη, στην Ιταλική ένομη τάξη είναι αδύνατον μία έρευνα να γίνει δηλαδή να, γίνουν, να γίνει παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών χωρίς να έχει δώσει άδεια ο εισαγγελέα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί η αστυνομία να, γίνει, να κάνει τέτοιου είδους έρευνες χωρίς να έχει την εντολή του δικαστή. Τώρα, το να αφαιρέσουμε από τον Ιταλό πολίτη το δικαίωμα να δίνει, να έχει την δικαστική εντολή, τη δικαστική ε, άδεια, αυτό είναι μια παραβίαση των δικαιωμάτων του. Τώρα, όσον αφορά τα ε, συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών εντάσσονται στα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα συντάγματα των κρατών μελών. Εγώ πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο ε, συλλάβαμε, αν θέλετε, αυτό το σχέδιο Ευρωπαϊκής ε, Εντολής Έρευνας είναι, έγινε με πάρα πολύ, πάρα πολύ βιαστικά, πραγματικά υπερβολικά βιαστικά πιστεύω, είναι καρπός μιας ε, έτσι πολύ γρήγορης ε, ε, αντιμετώπισης των πραγμάτων και μιας συνεργασίας των κρατών μελών χωρίς να έχει γίνει μια ενδελεχής μελέτη του θέματος. Ένα, μια ευρωπαϊκή εντολή έρευνας θα πρέπει να λειτουργεί μέσα σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια, δηλαδή να έχουμε τις συγκεκριμένες ποινικέ ε, ε, παραβιάσεις, ε, τα δικήματα δηλαδή, συγκεκριμένα δικαιώματα και συγκεκριμένα, συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Εδώ μιλάμε για όλα τα, τα δικήματα, για όλες τις μεθόδους. Δεν προβλέπεται δηλαδή μία έγκριση από πλευράς του εκτελούντος κράτους. Δηλαδή ακόμα και ο μηχανισμός ο οποίος προβλέπει από κάποια συντάγματα, θα μπορούσε θα μπορούσε να λειτουργήσει. Εδώ όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα προσεκτικά για να είμαστε σίγουροι, την κατάσταση, για να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, βέβαια γιατί θέλουμε να λειτουργήσει και να είναι αποτελεσματικός ο μηχανισμός, και θα πρέπει να εξεταστούν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Παραδείγματο χάρη η εντολή θα πρέπει να δίδεται από κάποιον συγκεκριμένο δικαστή όχι από οποιονδήποτε. Η εκτέλεση δεν θα είναι αυτόματη, αλλά θα πρέπει να εκδίδεται από κάποιον δικαστή και θα πρέπει να επικυρώνεται από τον δικαστή στην χώρα που θα εκτελεστεί η εντολή. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα προσφυγή σε έναν δικαστή της χώρας που εκτελεί το, την εντολή. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα. Δηλαδή, εάν ε, καλούμεθα να ερευνήσουμε ε, με, με βάση μια εντολή που προέρχεται από μια χώρα, αλλά στην χώρα εκτέλεσης ε, το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο έχει διαταχθεί η εντολή δεν αποτελεί αδίκημα, τι θα γίνει, πώς θα ερευνήσουμε για έναν πολίτη σε μια άλλη χώρα όπου σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία δεν έχει διαπράξει κανένα δίκημα. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει δηλαδή μια σειρά θεμάτων που θα πρέπει να εξετάσουμε, παραδείγματος χάρη. Ε, ο πολίτης πρέπει να σεβαστεί την νομοθεσία στην, ε, της χώρας στην οποία ε, ζει. Επομένως, όλα αυτά τα πράγματα δεν, δεν τα έχουμε διευκρινίσει. Ο κύριος Φως. Πριν επιστρέψουμε στον εισηγητή και στον οργανισμό. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά από όσα ήθελα να πω έχουν ήδη υποθεί και καλύφθηκα και θα περιοριστώ σε μία εκτίμηση και δύο παρατηρήσεις το, η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας θα μου φαινότανε πιο λογική αν είχαμε και κοινέ προδιαγραφέ στο ποινικό δίκαιο, στο σημείο 8 της ημερήσία ε, διάταξη, θα το συζητήσουμε και αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να συζητήσουμε πρώτα το 8 και μετά αυτό που λέμε τώρα. Εντάξει, τώρα το βάλαμε αλλιώ στην ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που είναι η προστασία των δεδομένων, ιδιαίτερα γιατί ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είπε ότι η απόφαση του 2008 δεν συμπεριλήφθη και το στυλίτευσε ίσως αυτό. Θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας στη διαβίβαση στοιχείων και δεδομένων και διασυνοριακά να γνωρίζουμε τι λέει και ο Οργανισμός ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να δίνουμε συνέχεια και να ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα αιτήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκριμ Χέντεν σημείωνε όλα αυτά που λέγατε και νομίζω καλό θα ήταν να του δώσουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσει πριν δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας κύριο Μέλο για να ολοκληρώσει. Η Προεδρία του Συμβουλίου μήπως θέλει να μιλήσει. Ωραία. Πριν τον κύριο Μέλο, αλλά πρώτο οργανισμός. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι κράτησα σημειώσεις κυρίως για μένα γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ένα σχόλιο μόνο που διατυπώθηκε ως ερώτημα και δεν μπορώ, έχω τον πειρασμό να απαντήσω. Έγινε αναφορά από τον κύριο Ντε Ιόγκ Ε, για να υπάρχει μία ρήτρα απόρριψη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και η κυρία Λάγκφορντ είπε ότι στη γνωμοδότηση πρέπει να τονίζουμε ότι θα υπάρχει ένας εύλογος, ένα εύλογο επιχείρημα ε, ίσως από τον τομέα του ασύλου ε, για να εφαρμοστεί αυτή η ρήτρα ή να υπάρχουν ορισμένα χρονικά περιθώρια ή να υπάρχουν συγκεκριμένε προδιαγραφές για το βάρος της απόδειξης ή ορισμένες εγγύησεις για να μην χρησιμοποιείται υπερβολικά αυτή η εντολή. Τέλος πάντων να διασφαλίσουμε ότι όλη η διαδικασία θα είναι ομαλή ε, ένομοι και ότι δεν γίνονται παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στο Συμβούλιο, ε, αν έχει κάτι να προσθέσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του Συμβουλίου το, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία των κρατών μελών συζητείται ευδελεχώς στο Συμβούλιο αυτή την εποχή και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον οργανισμό για την γνωμοδότηση του. Βεβαίως τα πράγματα έχουν εξελιχθεί μεταξύ και τώρα συζητάμε τους, τα επιχειρήματα προς, για την απόρριψη ε, όπως παραδείγματο χάρη τον ενδεχόμενο κίνδυνο παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων κλπ. Συζητάμε λοιπόν τα αίτια, του λόγου απόρριψη και θα επανέλθουμε όταν έχει συμφωνηθεί η άποψη του, του Συμβουλίου. Αλλά οποιαδήποτε ε, πρόταση για το σχέδιο αυτό θα είναι χρήσιμη. Ορισμένε από αυτέ τι διατάξει βεβαίω θα συζητηθούν σε πολιτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια αυτή τη προεδρία, αλλά θα είναι αδύνατο να έχουμε ένα τελικό κείμενο μέχρι τον Ιούλιο. Είναι ένα μακροπρόθεσμο, ε, μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια αυτή και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Ο Πρόεδρος, σα ευχαριστώ κύριε Ζόντρα, με πλευρά του Συμβουλίου. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, δίνω τον, τον λόγο στον κύριο Μέλο για να ολοκληρώσει το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολλούς λόγους όπως θα λέγαμε στη χώρα, μας, στη χώρα μου, στην Πορτογαλία το σχέδιο αυτό θα πρέπει ακόμα να ψηθεί, είναι ακόμα άψητο όπως λέμε. Χρειάζεται πολύ ε, ψήσιμο ακόμα για να ολοκληρωθεί τέλο πάντων αυτή η γνωμοδότηση. Βεβαίω με 27 κράτη-μέλη είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε μια ταχεία διαδικασία έτσι ώστε να, καλυφθούν και οι έρευνες ποινική ε, φύσεως. Αυτά τα αδικήματα πολλές φορές είναι διασυνοριακά ή εμπλέκονται ε, δια, ομάδες ε, ε, ε, ε, αδικοπραγούν εγκληματιών και χρειάζεται χρόνος για να συλλέξουμε όλες τις, τα στοιχεία, όλες τις αποδείξεις. Παρ' όλα αυτά πρέπει να, ενεργούμε, πρέπει να ενεργούμε γρήγορα, δεν λέω, αλλά χρειάζεται και προσοχή για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με, όλες, με όλα τα διαφορετικά δίκαια, με τις ποινικέ διατάξεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και με τις ε, μεθόδους συλλογής ε, αποδεικτικών στοιχείων. Υπάρχουν επίσης αδικήματα σε ορισμένε χώρες τα οποία ε, είναι ποινικά και σε άλλες δεν χαρακτηρίζονται ως ποινικά αδικήματα. Υπάρχουν λοιπόν μεταξύ των κρατών μελών μεγάλες διαφορές ακόμα και στο δικαστικό σώμα, στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Παραδείγματος χάρη συλλογή DNA ε, ε, υπάρχουν τελείως διαφορετικές διατάξεις ε, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ελλάδος, Γερμανίας, Πορτογαλίας για το DNA. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και πολλούς άλλους είναι πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί μια τέτοια οδηγία. Και σας ζητώ εξ αρχή συγγνώμη, αλλά πρέπει να πω ότι είναι τόσο ασαφή όλα αυτά τα οποία λέει η έκθεση, είναι τόσο συγκεχημένα. Παραδείγματο χάρη στα συμπεράσματα, λέει η έκθεση, λαμβάνοντα υπόψη τη το ενδεχόμενο μιας αναθεώρησης επί τη βάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει η εντολή αυτή να είναι πάρα πολύ σωστά καθορισμένη και όλος ο μηχανισμός αυτός να λειτουργεί επί τη βάση εγγύησεων και ορισμένες εγγύησεις πρέπει να υιοθετηθούν. Ωραία τα λέει, αλλά συγκεχημένα είναι όλα αυτά. Ποιες εγγύησεις και πώς. Γι' αυτό λοιπόν τονίζω ότι ως θέμα αρχή, υπάρχει ένα θέμα αρχής. Το θέμα αυτό της εντολής είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Πρέπει να προχωρήσουμε, εντάξει. Όμως το γεγονός ότι τα, τα, τα συστήματα της, ε, οι ποινικέ δικονομίες και κώδικες διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, μας δημιουργούν ε, δυσκολίες. Παραδείγματος χάρη, ένας Πορτογάλος δικαστής πρέπει να ασχοληθεί με μια υπόθεση η οποία συνέβη στη Μάλτα ε, και θέλει να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία που προέρχονται από την Ελλάδα ή από το μέρος όπου διαπράξει το αδίκημα όλη αυτή η διαδικασία ξεπερνάει τις αρμοδιότητες όσον αφορά τις, ε, ε, τις, δικαστικές του αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι ε, υποθέσεις ε, χρειάζονται χρόνο. Εν τω μεταξύ προσβλέπουμε μεγάλη χαρά στις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα έχω με τους κοιόδης εισηγητές. Αυτή θα είναι η πρώτη γνωμοδότηση που θα παρουσιάσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι και εύκολη, δεν μου θέσετε μια εύκολη, αλλά οπωσδήποτε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Μέλο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γκριμχέντεν για την έκθεσή του από πλευρά οργανισμού, Ευρωπαϊκού Οργανισμού και θα συνεργαστούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα και στο μέλλον βεβαίω, συχνά με, την με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Γεια σα, σα ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Υπάρχουν 7. Κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχό του να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και που ενδεχομένως διαθέτουν θεώρηση και δημιουργία μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου. Ε, Το σημείο αυτό έχει συγκίτρια την κυρία Τάνια Φανιχιών. για να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που να βεβαιώνει ότι τα έγγραφα, τα οποία ταξιδιωτικά έγγραφα έχουν εκδώσει τρίτες χώρες, είναι επίκαιρα και εγκαίρως ενημερωμένα. Η κυρία Φαγιόν θα μας παρουσιάσει τη έκθεση, το σχέδιο έκθεσης και μετά θα το συζητήσουμε με τα άλλα μέλη. Έχει το λόγο η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω και στους συναδέλφους ότι θα υποφεληθώ της παρουσίας των διερμηνέων και θα μιλήσω σλοβενικά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή Μάσα... Ε, προχωράει για την διαδικασία αυτή και μπορούμε σήμερα να ε, συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης το οποίο προετοιμάζω. Ε, συζήτησα το θέμα και με άλλους συζητητές ε, αλλά και με εκπροσώπους της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία. Η έκθεση αυτή είναι τεχνικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα όμως έχει και ένα συγκεκριμένο πολιτικό βάρος. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις σας. Η πρότασή μου δεν, δεν περιλαμβάνει πολλές τροπολογίες στην πρόταση της Κομισιόν. Η Κομισιόν στην πρόταση της προτείνει έναν μηχανισμό για την σύνταξη ενός καταλόγου ταξιδιωτικών εγγράφων με τα οποία μπορούν οι, οι, πολίτες να περνούν τα εξωτερικά σύνορα. Ανεπίσημα υπήρχαν τέτοιου είδου κατάλογοι, όμως τα κράτη-μέλη και, τα τρίτα, και τρίτες χώρες δεν είχαν ε, υποχρέωση να κοινοποιούν ε, την αναγνώριση, τη μη αναγνώριση ε, καινούριων ταξιδιωτικών εγγράφων. Και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εφόσον η πρόταση αυτή βέβαια ε, εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κατάσταση αυτή θα αλλάξει. Αυτός ο κατάλογος θα είναι νομικά δεσμευτικός και θα ε, είναι προσπελάσιμος, αν θέλετε, και στο ίντερνετ. Επίσης κάτι άλλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας ενημερώνει, το μας αφορά, θα μας αφορά για τις προτινόμενες αλλαγές και με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να αντιδρούμε στις προτινόμενες αλλαγές. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο ε, στην πρότασή μου που θα ήθελα να τονίσω. Η, προ... η Κομισιόν στην πρότασή της, στην πρόταση σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν ποια ταξιδιωτικά έγγραφα αναγνωρίζουν και ποια δεν αναγνωρίζουν, η Κομισιόν δεν Ευκρινίζει τι θα γίνει εάν μια χώρα δεν ε, κάνει την ε, κοινοποίηση μέσα σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Η πρότασή μου είναι ότι αν ένα κράτος μέλος δεν κοινοποιεί τη θέση της ε, σχετικά με ένα ταξιδιωτικό έγγραφο, αυτό σημαίνει αυτόματα την αναγνώριση του ταξιδιωτικού εγγράφου από το εν λόγω κράτος μέλος. Με τον τρόπο αυτό τα κράτη-μέλη θα έχουν και ένα κίνητρο για να δηλώνουν τις ε, θέσεις τους εγκαίρως και με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί και το ταξίδι των ε, πολιτών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στο παρελθόν είχαμε κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις ε, που οφείλονταν στο γεγονός ότι δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός για την ανανέωση και την προσαρμογή του καταλόγου. Πολλές φορές στα σύνορα κάποιοι αρνούνταν την είσοδο κάποιων πολιτών που είχαν κάποια ταξιδιωτικά έγγραφα διότι δεν γνώριζαν γνώριζαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή κάποιες χώρες για πολιτικούς λόγους δεν ενέκριναν ε, τα ταξιδιωτικά έγγραφα κάποιων χωρών. Παραδείγματο χάρη ε, ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδει το, κοσυφοπαίδιο. Δεν ε, μπορούμε να παρέμβουμε βέβαια στο κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών μελών να αναγνωρίζουν ή όχι κάποια ταξιδιωτικά έγγραφα. Δεν μιλάμε για την αναγνώριση, μιλάμε για την κοινοποίηση Τη αναγνώριση ή μη αναγνωρίση των, ε, των ταξιδιωτικών εγγράφων. Και τα κράτη-μέλη έχουν ε, μία δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίε για τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία αναγνωρίζουν ή δεν αναγνωρίζουν. Αυτό ε, αφορά επίσης και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση μιας επιτροπής. Επιτροπής που θα λειτουργεί σαν πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις στα σύνορα, θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιό να ε, ολοκληρώσει εδώ πιο γρήγορα μια ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων που θα επιτρέπει την ε, εμφάνιση οπτικά των ε, ταξιδιωτικών γράφων. Αυτό θα βοηθήσει περισσότερο τους, τελο, τους φρουρούς των συνόρων. διότι καλό θα είναι να έχουν ε, μία δυνατότητα οι, ε, φρουροί των συνόρων να ενημερώνονται online ε, και να βλέπουν οπτικά την, ε, τα κείμενα. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει, μέχρι ότου υλοποιηθεί η πρόταση αυτή. Θα ήθελα να σας ζητήσω επίσης ε, μέχρι τις 5 η ώρα την, ε, ε, Δευτέρα να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας γιατί αρχές Απριλίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και μετά ούτως ή άλλως την συνάντηση που είχαμε τους σκιώδεις εισηγητές δεν περιμένω οποιαδήποτε επιπλοκή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φαγιάν. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουν να πούν τα μέλη της Επιτροπής μας πρώτα. Η κυρία Νεντέλτσεβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της και για την εκτενέστατη παρουσίαση που μας έκανε τώρα. Χτες συνεδριάσαμε μαζί όλοι οι σκιώδεις συγητές. Ήταν αρκετά παραγωγική η συνεδρίαση ομολογώ και γενικά δεν έχουμε μεγάλες ε, διαφορές. Ήταν μια συνεδρίαση που μας επέτρεψε να διευκρινίσουμε περισσότερο τα πράγματα και να υποστηρίξουμε κάποιες θέσεις που θέλουμε εδώ στο Κοινοβούλιο να υποστηρίξουμε. Εγώ είχα δύο ερωτηματικά. Και τα δύο απαντήθηκαν χτε μετά από τη συνάντηση αυτή που είχαμε πραγματικά καρποφόρα. Ε, η πρώτη μου ανησυχία και μέλημα ήταν ποιο θα είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτέ τι διαδικασίε. Αλλά η κυρία Φαγιόν μου είπε ότι θα κάνει τεχνικέ τροπολογίε σχετικά με του νέου κανόνε για την επιτροπολογία, οπότε μα διαβεβαιώνει ότι θα ακολουθήσει ε, αυτού του κανόνε και το Κοινοβούλιο. Και η δεύτερη ανησυχία μου αφορούσε τη δυνατότητα να είναι πιο αποτελεσματική η έλεγχη και στα εξωτερικά σύνορα αλλά και ε, από το προσωπικό των προξενικών αρχών. Και ε, ρωτώ, τι δυνατότητες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να θέσει στη διάθεση των κρατών μελών μια ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων για όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα που αναγνωρίζουν τα κράτη-μέλη. Λέει η συγκήτρια ότι αυτό θα γίνει, ε, επίκειται, ας ελπίσουμε να γίνει σύντομα. Σε ό,τι αφορά τώρα την προθεσμία που θα έχουν τα κράτη-μέλη για να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναγνώριση ή μη αναγνώριση των εγγράφων και αυτή τη στιγμή παρέλθει αυτή η προθεσμία, θεωρείται αυτόματη αναγνώριση, υποστηρίζω την εισηγήτρια και θέλω να την ευχαριστήσω και πάλι για τη συνεργασία και για την πολύ καλή δουλειά της. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ο κύριος Ταβάρες Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο εγώ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φαγιόν και εγώ με τη σειρά μου για τη συνεργασία που είχαμε. Και για την προθυμία που είχε πάντα να ε, δέχεται ε, προτάσεις και είναι και ίδια πάρα πολύ ε, συνεργάσιμη. συμφωνώ με την ιδέα αυτή να έχουμε ε, υποδείγματα ε, ταξιδιωτικών εγγράφων σε μία βάση δεδομένων. Ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό για τους υπαλλήλους για να αναγνωρίζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Στα εξωτερικά σύνορα για πολίτες των τρίτων χωρών της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται στο εσωτερικό της Ένωσης. αλλά έχω λάβει πολλές καταγγελίες και παράπονα από πολίτες της δικής μου χώρας. Όταν αλλάζουμε κάτι στα ταξιδιωτικά μας έγγραφα, τις ταυτότητες, τα διαβατήρια, υπάρχουν χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν θεωρούν έγκυρα αυτά τα έγγραφα, γιατί δεν τα ξέρουν, δεν τα αναγνωρίζουν. Ε, εντός και εκτός του Σέγγεν. Είναι καλό αυτό λοιπόν για τα εξωτερικά σύνορα, νομίζω θα ε, έπρεπε να το επεκτείνουμε σε όλα τα κράτη-μέλη, για να βεβαιωνόμαστε ότι και οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα. Και στη συνέχεια υποστηρίζουμε χωρίς καμία επιφύλαξη την ιδέα αυτή ότι η προθεσμία του ενός μηνός αρκεί ε, για να ε, εγκρίνουν ή να απορρίπτουν τη θεώρηση διαβατηρίου τα κράτη-μέλη και από εκεί και πέρα ε, θα μπορούμε να εγκρίνουμε ε, τη θεώρηση από την παρέλευση ενός μηνός και μετά. Και επίσης όταν υπάρχει απόρριψη, άρνηση από ένα κράτος μέλος, χρειάζεται λεπτομερή αιτιολόγηση. Αυτές είναι τρεις ιδέες για μας σημαντικές και μπαίνουν και στην έκθεση της κυρίας Φαγιών. Ευχαριστώ πολύ και ε, συμφωνούμε μαζί της. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Στάνοκα. Yes, ε, thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ μαζί με τους άλλους συναδέλφους. Θα ήθελα να σε χαρώ την κυρία Φαζόν για την εργασία της αυτή και ε, στις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών βεβαιώσαμε πολλά στοιχεία. Δεν νομίζω να υπάρξουν προβλήματα στην εξέλιξη. Ε, τροπολογίες θα υποβληθούν. Έχω την πρόθεση να υποβάλω μερικές τροπολογίες το έγγραφο δεν αναφέρει ότι πάνω από 15% του πλουσισμού της Λετωνίας, της χώρας μου, έχουν παραλυφθεί από το έγγραφο αυτό, το οποίο προετοιμάστηκε από το Συμβούλιο, συντάχθηκε από το Συμβούλιο και δυστυχώς και οι αρχές παρέλειψαν να το πράξουν της χώρας μου είναι ένα ειδικό καθεστώς όπως έχει καθοριστεί συνταγματικά από πολίτες που δεν είναι πολίτες της Λετωνίας, άνθρωποι που δεν είναι πολίτες, αλλά είναι απάτριδες. Έχουν ένα ειδικό καθεστώς πρώην πολιτών της ε, ΕΣΔ, της ε, Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, είναι λοιπόν μια ειδική ομάδα αυτή και ε, οι διαδικασίες που ισχύουν για τις θεωρήσεις ισχύουν και για αυτούς, δηλαδή πολίτες που είναι πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής άνθρωποι που δεν είναι ε, ε, Ευρωπαίοι, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και απάτριδες πρέπει να επαχθούν σε κάποιο καθεστώς θεωρήσεων. Ελπίζω αυτό το 15% του πληθυσμού μας να μην ξεχαστεί τελείως και να βρεθεί κάποια λύση και σας υπενθυμίζω επίσης ότι είχαμε μια πρόθεση να οργανώσουμε μια κρόαση για αυτούς τους ανθρώπους του ειδικού καθεστώτος. Yes. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Στάνο, καλή ο πρόεδρος. Θα ήθελε άλλο συνάδελφο να λάβει το λόγο, όχι. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Προεδρία. Η Κομισιόν εκπροσωπείται από τον κύριο Γιάννη Ντεκώστε. Θέλετε το λόγο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα προς συζήτηση. Πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες που ήδη έχει προτείνει είναι αποδεκτές ε, για μας Ιδιαίτερα η τρίτη τροπολογία που προσπαθεί να συμπληρώσει ένα νομικό κενό στο τρέχον σύστημα, δηλαδή να καθορίσουμε τι θα γίνει αν το κράτος μέλος δεν λάβει απόφαση, αν θα αναγνωρίσει ή όχι ένα συγκεκριμένο τεξιδιτικό έγγραφο. Την ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την τροπολογία τρία και αυτή θα ενισχύσει βεβαίως και τη θέση ε, στο Συμβούλιο ε, πολύ. ορισμενα ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να μην δεχτούν μια τέτοια λύση, αλλά εμεί συμφωνούμε. Όσον αφορά το σχόλιο για τους απάτριδες που ζουν στη Λετωνία, εδώ μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ε, σύμφωνα με την αρχική πρόθεση της Κομισιόν που είναι να καλύψει όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα που δίδονται, που παρέχονται σε υπηκόους τρίτων χωρών, δηλαδή όχι Ευρωπα... Ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τα άτομα αυτά τα οποία δεν λαμβάνουν τα, τα έγγραφα για τους απάτριδες από τη Σύμβαση του 1954, τα άτομα αυτά δεν θα ξεχαστούν. Το Συμβούλιο σκέφτεται, αναλογίζεται αυτή την ειδική κατάσταση και η Κομισιόν δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να καλυφθεί και αυτή η περίπτωση. Τελευταία παρατήρηση είναι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων και το δείγμα. Με το δείγμα Όπω είπαμε, όταν για πρώτη φορά συζητήσαμε αυτή την πρόταση της, Κομισι... Κομισιόν, δεν... Της, επιτροπής, επιτροπής αυτής. Δεν έχουμε πρόβλημα το να δεχτούμε τη σύσταση ε, μιας τέτοιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όμως είναι ε, επίγον να διορθώσουμε, να βελτιώσουμε το τρέχον δυσλειτουργικό σύστημα που έχουμε ε, και ελπίζω σύντομα όχι μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να το επιτύχουμε. Διότι ε, δέχεται να καθυστερήσει η υιοθέτηση αυτού του μέσου, το οποίο ε, νομικό μέσον αυτό πρέπει να επικυρωθεί, να υιοθετηθεί για να λυθούν τα τρέχοντα προβλήματα. Θα υπάρχει λοιπόν μια τροπολογία επί του στο πρωινή, στο εκτιμώντας, που θα προτείνει την ε, εφαρμογή αυτής της ιδέας, ε, την, μεταφορά αυτής της ιδέας σε, πρακτική εφαρμογή. Ε, άρα αυτό λοιπόν είναι μία προϋπόθεση για μας να λυθεί αυτό το πρόβλημα προηγουμένως πριν υιοθετηθεί αυτή η πρόταση. Ο Ευχαριστώ. Από το Συμβούλιο, ο κύριος Σόργη, παρακαλώ. Θέλει επίση το λόγο να πει τίποτα. Ορίστε. Eh, Ευχαριστώ. Συντομία να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Να ευχαριστήσω την κυρία Ταχών καταρχάς για, την, για το σχέδιο έκθεσής της. Πρέπει να πω ότι το περιεχόμενο της έκθεσης έχει συζητηθεί στην ε, ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για, την, ε, για τις άδειες διάλευσης, για, τις, για την βίζα, γιατί είναι η ομάδα που είναι υπεύθυνη και θα, θα συνεδριάσει και αύριο για να συζητήσει το σχέδιο πρότασης. Ε, η, η έκθεση της κυρίας Φαγών ευθυγραμμίζεται ε, απόλυτα και με, την, ε, με τις θέσεις των κρατών μελών. Βρίσκει σύμφωνο η γνωμοδότηση αυτή την, το Συμβούλιο για το άρθρο 4 δηλαδή για, το, για την περίπτωση που δεν ε, ανακοινώσει ένα κράτος μέλος την άποψή του για κάποιο ταξιδιωτικό έγγραφο, θα πρέπει αυτόματα να θεωρήσουμε ότι δεν το αναγνωρίζει. Αυτή είναι μια άποψη την οποία δεν δέχονται τα, όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και, το, η Προεδρία. Κάτι αντίστοιχο έχει προτείνει και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια συνένεση σε επίπεδο ομάδας Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Το λόγο ξανά τώρα η συγγήτρια Τάνια Φαγιών για να ολοκληρώσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για την ενημέρωση, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και τους σκιώδης ηγητές. Γενικά βλέπω ότι είναι κοινή η αίσθηση και η συμφωνία μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα τέτοιο μηχανισμό. Θα επιθυμούσα πάρα πολύ η πρωτοβουλία αυτή να βρει και τη συμφωνία του Συμβουλίου. Δηλαδή ότι ένα κράτος που δεν θα έχει αποφανθεί εντός του μηνός θα θεωρείται ότι το αναγνωρίζει και ελπίζω αυτό να εγκριθεί ομόφωνα στο Συμβούλιο. Ελπίζω να έχουμε και νομίζω ότι έχουμε την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων προς τα εκεί και επίσης θα ήθελα να συμβουλεύσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το σκεφτεί αυτό το θέμα της Τράπεζας Δεδομένων μακροπρόθεσμα, δεν λέω τώρα, για να ε, υπάρχει και αυτό το υλικό, φωτογραφίες με τα δείγματα των ταξιδιωτικών ε, εγγράφων, είναι σημαντικό. Και ο κύριος Σταβάρης είπε κάτι για κάποια εικονικά ταξιδιωτικά έγγραφα. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει αφήσει εκτός της πρότασης, γιατί ε, για μένα δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος να μπει, δεν έχει προστιθέμενη αξία. Δεν ξέρω αν θέλουμε για το μέλλον να κάνουμε ένα τέτοιο κατάλογο, να ξέρουν οι, οι μεθοριακές αρχές τι ε, υπάρχει και αν τυχόν ε, υπάρχουν εικονικά ή πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα να τα έχουν και αυτά υπόψη του. Εγώ δεν ξέρω στο παρελθόν τι εμπειρία νομίζω ε, δεν είχαμε. Για την επιτροπολογία, τα είπα και χτες, στη συνάντηση με τους ε, σκιώδει εισηγητές. Θα πρέπει να τηρηθούν κάποιε διαδικασίε σύμφωνα με τη νέα πλέον μέθοδο που ακολουθούμε τη συνθήκη της Λισαβόνας για να μην έχουμε εκπλήξεις. Νομίζω είναι 7 οι ε, συμπληρώσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει έτσι κι τη δυνατότητα να αποφαίνεται για κάθε αλλαγή. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να μας στείλει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κάθε φορά που αλλάζει ένα έγγραφο που αναγνωρίζεται ή δεν αναγνωρίζεται. Λοιπόν, λαμβάνω υπόψη μου όλα αυτά που είπατε και θα περιμένω και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και για την προθυμία σας, κυρία Φαγιόν και το ανοιχτό πνεύμα με το οποίο εξετάζετε τις προτάσεις των συναδελφών. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να περάσουμε για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα στην εξή ανακοίνωση. ημέρα Δευτέρα κατάθεση τροπολογιών. 21η Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα. 5 ώρα το απόγευμα. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 12 Απριλίου στην Επιτροπή μας. Εντάξει, συμφωνείτε. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα εδώ και προχωρούμε στο επόμενο. Έχουμε ακόμα και συντονιστές. Μην ξεχνάτε, 6 με 6,5. Έχουμε όμως και άλλο θέμα ενδιαφέρον, το 8. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων είναι για την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Γνωρίζετε ότι λόγω της σημασίας τη ποινική δικαιοσύνης μετά τη θέση σε ισχύ της Ειδικής αγώνα. οι συντονιστές ε, της Επιτροπής μας αποφάσισαν να αφιερώσουν μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία στο ποινικό δίκαιο. Ο τίτλος της έκθεσης άλλαξε και είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ποινικό δίκαιο. Σήμερα θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα αυτά και θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας, κύριο Ντογιόγκ. Μπορεί να μας παρουσιάσει λοιπόν τις απόψεις του. Μετά μπορεί να θέλει μιλήσει και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι συνάδελφοι. Mr. De Jong, as rapporteur, you got the floor. Ο κύριος De Jong, εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφέρατε τον τίτλο διότι στην ημερήσια διάταξη λέει ακόμα εναρμόνιση του ποινικού δικαίου και τώρα αποφάσισαν οι συντονιστέ να χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ποινικού δικαίου. Όσον αφορά τη διαδικασία, έχω δώσει στη γραμματεία ένα σχέδιο για τη συζήτηση σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζω να έχει διανεμηθεί αυτή η σκιαγράφηση πρώτη της συζήτησης που περιλαμβάνει τα πιο ουσιαστικά σημεία. Δεύτερον, θα ήθελα να ξέρω εάν οι σκιώδεις εισηγητές για αυτή τη γνωμοδότηση ενδιαφέρονται να οργανώσουμε μία συνάντηση πριν υποβάλω το σχέδιο έκθεσης. Εάν, ναι, αν ενδιαφέρονται, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις διάφορες ιδέες μας σε πιο πολλές λεπτομέρειες πριν ολοκληρώσω το σχέδιο, τη σύνταξη του σχεδίου γνωμοδότησης. Τώρα η ουσία. Ο στόχος της έκθεσης αυτής, η από ό,τι αποφασίστηκε ή συζήτησαν οι συντονιστές είναι το ποινικό δίκαιο Uh, Το εμπράγματο. Το εμπράγματο ποινικό δίκαιο. Και ε, ξέρουμε ε, από προηγούμενες εκθέσεις του Κοινοβουλίου ε, ότι έχουν γίνει γνωμοδοτήσεις για άλλες πτυχές του ποινικού δικαίου. Δεύτερον, γιατί τώρα εστιάζουμε στο εμπράγματο γιατί το ποινικό δίκαιο έχει δύο πτυχές. Από τη μία πλευρά είναι συνήθως η απάντηση σε πολιτικό επίπεδο, όταν ένα πρόβλημα προκύψει και για, όταν θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε δραστήριοι και κάνουμε κάτι, αμέσως αναφερόμαστε στο ποινικό δίκαιο, ενώ στο, στην, ε, όσον αφορά το το, κοινοτικό δίκαιο. Α, όχι. Όσον αφορά δε το ποινικό κώδικα, ε, ε, συνήθως προκύπτει θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν καταφεύγουμε στον ποινικό, στην ποινική δικονομία πολλές φορές ε, υπησέρχονται θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά άλογα με το πώς εφαρμόζεται το, το ποινικό δίκαιο στα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν πρέπει από τη μία πλευρά να έχουμε υπόψη μας την ευρωπαϊκή νομοθεσία της Ένωσης δηλαδή και από την άλλη να ξέρουμε τις επιπτώσεις τους ανάλογα με τα ποινικά δίκαια των διαφόρων κρατών μελών. Αυτό το άρθρο 83 της συνθήκης της Ένωσης επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη και επίσης το 2009 το Συμβούλιο είχε υιοθετήσει συμπεράσματα και διατάξεις όσον αφορά τις διαβουλεύσεις του Συμβουλίου για το ποινικό δίκαιο. Ορισμένα από τα κείμενα τα οποία υιοθέτησε τότε το, το Συμβούλιο είναι πολύ ενδιαφέροντα, όμως από διαδικαστική άποψη είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Πριν ισχύσει η συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε τη δυνατότητα να τα συζητήσει και η Κομισιό κράτησε απόσταση από αυτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και έκανε μια δική της ξεχωριστή ε, δήλωση. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να ξέρουμε ποια ακριβώς είναι η θέση αυτών των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το ποινικό δίκαιο. Πρέπει όμως να το κάνουμε αυτό με την συμμετοχή της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να δούμε που, πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση μετά τα συμπεράσματα. Εξέτασα λοιπόν όσον αφορά τη γνωμοδότηση ε, το σύστημα στις Ηνωμένε Πολιτείες με πιστεύοντας ότι μπορούμε να μάθουμε κάτι και δεδομένου ότι έχουν μια ομοσπονδιακή νομοθεσία και ε, πολιτιακή νομοθεσία, μήπως μπορούμε να μάθουμε και να μας χρησιμεύσουν διάφορα στοιχεία. Δεν νομίζω όμως ότι τα πράγματα, ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη εμπειρία η αμερικανική, μάλλον αρνητική είναι. Δεύτερον, βάσει της συνθήκης και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να ε, αποφασίσουμε διάφορα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ισχύουν. Αυτά πρώτο, το πρώτο μέρος της γνωμοδότησης. Το δεύτερο αφορά το ποιοτικό στοιχείο του ποινικού δικαίου. Έχουμε στο, στο ποινικό ποινικό δίκαιο, ε, διάφορα στοιχεία τα οποία βασίζονται στο, στο ποινικό δίκαιο και αν έχουν επίπτωση στη φύση των διατάξεων. Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο στην αξιολόγηση των μέσων εφαρμογής του ποινικού δικαίου. Θα είναι πολύ χρήσιμο για το Κοινοβούλιο να αποφασίσει μία δέσμη αρχών, βασικών αρχών, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν, διάφορες, ε, υπάρχουν αρχές, συγκεκριμένες αρχές, κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Στεμελιώδεις αρχές μάλλον που πρέπει να ισχύουν το τρίτο μέρος της έκθεσης θα αφιερωθεί στις ε, θεσμικές ε, ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, διότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα σε όλα τα ευρωπαϊκά στους όλους θεσμικά όργανα που να ισχύσει ε, αυτή η προσέγγιση. Δεν ξέρω δεν γνωρίζω να υπάρχει κανένα σύστημα επί το οποίο έχουν συμφωνήσει όλα τα κράτη-μέλη, ούτε στο Συμβούλιο, ούτε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε ποτέ τη φιλοδοξία να χειριστούμε όλες τις προτάσεις όλων των διαφορετικών ποινικών ε, δικαίων ε, και να τα ε, εναρμονίσουμε ή να ακολουθήσουμε μία νέα προσέγγιση, αλλά είναι σημαντικό, και εδώ έχω υπόψη μου τις νομικές υπηρεσίες του σώματος, να πούμε ότι εγώ θέλω να είναι συνεκτικό το ποινικό δίκαιο, να υπάρχει συνοχή και ε, να ε, δούμε πώς μπορεί αυτή η συνοχή να εγγυηθεί, να, την, να εγγυηθούμε αυτή τη συνοχή από τις αρχές τις οποίες θα υιοθετήσουμε. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσω την άποψη και των άλλων συναδέλφων και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις που θα έχετε συγκεκριμένε. Ευχαριστώ κύριε Δεγιόγκ. Τώρα, όπως σας είπα, μπορεί να θέλουν να μιλήσουν βουλευτές, αλλά και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. από το Συμβούλιο, ο κύριος Πίτερ Σόγκα. θέλει να πει τίποτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί λαμβάνει η χώρα αυτή η συζήτηση τώρα που συζητάμε διάφορες προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου και πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο και μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης από το ε, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και κυρίως αναφορά και, και πιστεύω την και ε, θέματα που αφορούν το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονομία και θα πρέπει να υπάρξει μια συνέπεια ε, στις, στα μέτρα τα οποία υιοθετούμε. Αναφερθήκατε στις κατευθυντήρες γραμμές του Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν το 2009 ε, Υπάρχει και μια άλλη σειρά κατευθυντηρίων ε, γραμμών που υιοθετήθηκαν πριν από το 2009 και το Συμβούλιο σέβεται αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και τη σεβάστηκε και στο, σε επίπεδο εγγράφου το οποίο έγινε δεκτό από το Συμβούλιο, δηλαδή και την αρχή της αναλογικότητας και όσον αφορά την κλίμακα των κυρώσεων και των ποινών που αναφέρονται με λεπτομέρειες κατευθυντήρες γραμμές τις, όχι μόνο τις λάβουμε υπόψη μας, αλλά σεβόμαστε και κάποιες θεμελιώδεις αρχές ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνάμε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για την ένωση έτσι ώστε να ρυθμίζονται κάποια θέματα. Επομένως, αφήνουμε αρκετό, αρκετή ελευθερία στα κράτη-μέλη για να ρυθμίσουν τα θέματα αυτά, ε, σεβόμενοι την αρχή της επικουρκότητας. Επομένως, υπάρχει μια πολύ προσεκτική ισορροπία ε, για κάθε ε, πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Επομένω, αυτέ οι, οι κατευθυντήριε γραμμέ είναι μια ζωντανή πηγή έμπνευση για το Συμβούλιο όταν νομοθετεί. Αλλά βέβαια δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στο Συμβούλιο. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχει και μια σειρά αρχών που να γίνονται σεβαστές, να γίνονται σεβαστές από όλου. Και χαίρομαι γιατί το Συμβούλιο, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο κάθισε γύρω από ένα τραπέζι και συζήτησε όλα αυτά τα θέματα. Αυτή ήταν η βασική αρχή. Θα το θυμόσατε ότι και στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης υπήρχε μια γραμμή ότι όντω και αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ε, αντιμετώπιση τα τρία θεσμικά όργανα και ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα υποβάλει κάποιες προτάσεις βάσει των οποίων θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εν τω μεταξύ πιστεύω ότι ε, ασκείται μια πολιτική πολιτικού ποινικού δικαίου ε, κάθε μέρα. Ε, μιλάμε για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, ε, για την ε, ε, παράνομη διακίνηση παιδιών, ανθρώπων γενικότερα. Μέσα στα πλαίσια του τριλόγου ούτως ή άλλως εφαρμόζουμε την, τις κατευθυντήριες γραμμές. Τις κατευθυντήριες γραμμές που από το 2009 το Συμβούλιο εφαρμόζει. Μάλιστα. Α, έχουμε και μέλη που θέλουν το λόγο. Και η κυρία Λάτσφορτ και ο κύριος Γιακολίνο και ο κύριος Βό, άλλο. μόνο ένα πολύ. Λοιπόν, πρώτος ο κύριος Γιακολίνο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, πρόεδρε. Άκουσα τον εισηγητή και τους άλλους ομιλητές. Προφανώς θα άλλαζα και εγώ τον τίτλο αυτού του φακέλου. Θα έλεγα μία προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ποινικό δίκαιο. Και είναι πιο πολύ προσανατολισμοί θα έλεγα ότι είναι προσανατολισμοί που δημιουργήθηκαν μετά τη συνθήκη της, ε, της Λισαβόνας με βάση το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης. Είναι θέμα βέβαια εθνικής κυριαρχίας ε, το, το ποινικό δίκαιο. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τη τον διασυνοριακό χαρακτήρα της, του εγκλήματος, το, η διαπαρανομή διακίνηση ανθρώπων, ε, το ξέπλυμα του χρήματος κτλ. Επομένως, ε, μας αναγκάζουν να ε, αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας. Και πιστεύω ότι μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να, να συνδεθεί, αν θέλετε, και με μια πιο στενή συνεργασία ε, αυτών, αυτών που υπηρετούν ε, την, ε, τη δικαστική εξουσία. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μία εναρμόνιση του ποινικού δικαίου εάν δεν συνεργαστούν πιο στενά και οι δικαστές και όλοι όσοι ασχολούνται και όλοι όσοι ανήκουν στην δικαστική εξουσία. Γι' αυτό θα ακούσω με ιδιαίτερη προσοχή την συζήτηση που θα ακολουθήσει, θεωρώντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντική μια προσέγγιση που θα λάβει υπόψη την εφαρμογή του ποινικού δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη, οδηγώντας το σε μία προσέγγιση και διασφαλίζοντας και μάλλον και εξαγγέλλοντας την θέληση του Συμβουλίου να υπάρξει μια πιο στενή συνεργασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περνάμε μια πολύ ευαίσθητη πολιτική και ιστορική φάση. Ευχαριστώ. Η Λέδη Λάτφορντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σάρα, Σάρα, το, ο τίτλος μου δεν, έχει, δεν πειράζει. Είναι πραγματικά μια πολύ χρήσιμη άσκηση αυτή και θα έλεγα χωρίς αυτή την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας δεν θα είχα βρει και διαβάσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το ποινικό δίκαιο του 2009, οπότε είμαι πολύ ευγνώμων που βρήκα αυτά τα συμπεράσματα. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή ε, ε, κάθε φορά που χειριζόμαστε θέματα ποινικού δικαίου, ουσιαστικά ε, το εμπράγματο δίκαιο, και θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε αν υπάρχει μία συμβουλευτική υπηρεσία μέσα στη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου με στόχο την βελτίωση της νομοθεσίας. Ε, δηλαδή, εγώ θα ήθελα να έχουμε νομικούς εμπειρογνώμονες ε, να μας βοηθήσουν στη σύνταξη αυτών των ε, κειμένων, διότι πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είμαστε πολλοί ερασιτέχνε. ενεργούμε σαν ερασιτέχνε. Δεν είμαστε ούτε δικηγόροι, ούτε νομικοί, ούτε εμπειρογνώμονες σε αυτά τα θέματα, αλλά είμαστε νομοθέτες. Και θα πρέπει να προσέξουμε το κύρος μας ε, ε, έναντι των πολιτών της Ένωσης. Πρέπει όλα αυτά τα κείμενα νομοθετικού περιεχομένου να έχουν συνταχθεί με εξαιρετική προσοχή και να είναι ακριβέστατα. Επίσης, η επικουρικότητα, η αναλογικότητα, όλες αυτές οι αρχές πρέπει να γίνουν σεβαστές και να υπάρχει και πρόσθετη αξία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε θέματα που άπτονται του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που έγινε, που ανέφερε ο κύριος Ζόνκερ, ο κύριος Ζόνκερ, Ζόνκερ, ο πρόεδρος ε, του Συμβουλίου την ε, ιδέα αυτή της ε, πρόωθησης του θέματος και την ιδέα μιας τριμερούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο οπωσδήποτε μπορεί να αποφεληθεί από αυτό το μοντέλο που παρουσιάζει που, το μοντέλο που παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009. Στόχος μας είναι πάντοτε η βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας μας. Όσον αφορά τώρα στα ε, σχόλια του κυρίου Ζόγκα και όταν εγώ έκανα την εισήγηση πέρσι για τα θέματα τα διερμηνίες και μετάφρασης πέρσι ε, ε, πρέπει να εξετάσω λεπτομερώς το κείμενο διότι έχω ένα σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου που λέει ότι η Κομισιόν θα υποβάλει μια δήλωση που θα περιληφθεί στα πρακτικά. Ε, έτσι λέει το κείμενο του Συμβουλίου και πρέπει να βρω ήταν, ποια ήταν αυτή η δήλωση της Κομισιόν και τι λέει. Εν πάση περιπτώσει θα κάνω ό,τι μπορώ και θα συνεργαστώ με τον εισηγητή κύριο De Jong για αυτό το θέμα και είναι σωστό ότι χρειάζεται πειθαρχία και δεν μπορούμε έτσι στο γόνατο να πάρουμε αποφάσεις ε, που έχουν επιπτώσει στην ποινική δικονομία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η έκθεση θα μας οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση. Bene. Axel Ο κύριος Άξελ ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω ε, κύριε Ντε για την έκθεση αυτή. Ε, ασχολείστε πάρα πολύ εντατικά και κατά την άποψή μου θα πρέπει να ε, το προωθήσουμε και εμείς με φιλοδοξία και αυτό που είπε και η Σάρα να το λάβουμε επίσης υπόψη, ότι το εθνικό ποινικό δίκαιο είναι κάτι το οποίο έχει αναπτυχθεί για τη σειρά των αιώνων. Ε, και τη διάρκεια των αιώνων και έχουν και ιδιαιτερότητες στις χώρες τα εθνικά ποινικά δίκαια και θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο γίνεται, ε, έτσι, διαφυλάσσοντας και τα συμφέροντα αυτά, να προχωρούμε. Γενικότερα, θα ήθελα να πω ούτως ή άλλως απορροφούμε διάφορες ε, ε, αλλαγές που γίνονται σε άλλα συστήματα. Δεν υπάρχει ένα κλειστό σύστημα. Προφανώς και η νομολογία μας ε, και η νομοθεσία μας λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε άλλα νομικά συστήματα. Το να πιέσουμε όμως την κατάσταση νομίζω ότι δεν θα είναι ε, καλό. Και θα υπάρχει, θα δημιουργηθεί μια αντίσταση, αν θέλετε, ακόμα και στις απαραίτητες αλλαγές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η Προεδρία, η Ουγγρική Προεδρία θέλει να προσθέσει κάτι. Mr. Chairman, uh, Κύριε Πρόεδρε, απλώς θα να επαναλάβω αυτό που ήδη είπα. Ε, χαιρετίζουμε αυτή την πρώτη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα η ε, συμπερίληψη αυτών των πολύ καλών αρχών σε ένα ε, κείμενο ε, της Κομισιόν και του Συμβουλίου ή ενδεχομένως σε κάποια διαθεσμική μορφή. Και καλό θα ήταν να συζητήσουμε άτυπα, να κάνουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε αυτό το θέμα άτυπα. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Και εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Η Κομισιόν πιστεύει ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το νομικό τοπίο έχει μετα... αλλάξει πάρα πολύ, έχει μεταβληθεί μετά τη Λισαβόνα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις στα θεσμικά όργανα, αλλά επιτέλους πρέπει να σκεφτούμε με μια οριζόντια προσέγγιση και να σκεφτούμε το μελλοντικό πλαίσιο. Το κείμενο της, μέσα στην Κομισιόν ε, γίνονται πολύ σοβαρές συζητήσεις ε, ε, στις διάφορες υπηρεσίες και μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Οι γενικές διευθύνσεις εξετάζουν τυχόν προτάσεις, διατάξεις νομικές και από τη στιγμή, δεδομένου ότι έχουμε τώρα και την Γενική Διεύθυνση Λέξη, έχουμε συγκεκριμένη υπηρεσία για το ποινικό δίκαιο, ουσιαστικό και δικονομία και γι' αυτό θέλουμε ακριβώς να εργαστούμε για την επίτευξη μιας καλύτερης ε, συνέπειας, μια, μιας συνεπούς νομοθεσίας, ε, η οποία να ορίζεται από το στοιχείο της συνέπειας. Ευχαριστώ για την Κομισιόν και δίνω το λόγο τώρα στον ε, εισηγητή, τον κύριο Ντεγιόγκ, για, να, για, την πρώτη, για τα πρώτα συμπεράσματα από αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ε, ε, ακούσαμε τις αντιδράσεις των συναδέλφων του Συμβουλίου και της Κομισιόν και οι πρώτες αυτές αντιδράσεις ε, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να κάνουμε και άλλη μια συνάντηση πριν αρχίσουμε να συντάσσουμε το κείμενο και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, λάβει χώρα αυτή η συνάντηση. Θα πρέπει να συμφωνήσει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Τέλος πάντων, υπάρχει μία διαφορά σε σχέση με αυτά τα οποία ε, είπα στην αρχή για την ποινική δικονομία υπάρχει μια έκθεση του 2007 από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και εκεί με αυτή την έκθεση κανείς δεν είχε καμία αντίρρηση. Τώρα, αν θέλετε να το, να διευρύνουμε και αν θέλετε να ακολουθήσουμε τις προτάσεις του κ. Φως, δεν έχω καμία αντίρρηση να το κάνω. Ευχαριστώ. Με την παρέμβαση αυτή του εισηγητή, Α, όχι. Υπάρχει. Υπάρχει κι άλλη μια παρατήρηση. Η κυρία Λάντφοιντ. Βλέποντας το site του BBC για, τις, ε, για τα προβλήματα της λειτουργίας ε, ε, του, της Europol, να σας πω ότι ο κύριος Βουέν Ράιτα έδισε, έδινε μία συνέντευξη όπου έλεγε ότι ε, εξαρθρώθηκε το μεγαλύτερο δίκτυο παιδεραστίας που είχε ε, ε, βρεθεί ποτέ. Επομένως ο κύριος Wainwright έκανε τη δουλειά για την οποία να πληρώνεται, δηλαδή έκανε τη δουλειά της Europol. Τώρα αν αυτό τον ε, το να παλάσει από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση προς εμάς, αυτό είναι άλλη μια ιστορία. Λοιπόν, μετά από αυτά που είπε η Βαρονέσα, νομίζω ότι, η Βαρόνη, συγγνώμη, νομίζω ότι μπορούμε να διακόψουμε και δίνουμε ραντεβού αύριο στις 9. Θα γίνει μια πρώτη συνάντηση κυκλισμένων των θυρών με την ε, Επίτροπο την κυρία Μάλστρουμ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεδριάσουν οι συντονιστές σε λίγα λεπτά.